Ξεκινούμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Δεν έχει έρθει ακόμη συνάδελφοι από το ΕΛΚ γιατί έχουν άλλη συνεδρίαση παράλληλα, αλλά φαντάζομαι θα καταφτάσουν εντό ολίγου. Όπως ξέρετε και θα διαβάσετε και στο πρόγραμμά μας, θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση του κυρίου Κρίς Μπότερμαν που θα μας παρουσιάσει την έκθεση της Αγκαιόπα για το κοινωνικό διάλογο ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού dumping και της αδήλωτης εργασίας στη Γεωργία. Η έκθεση εκπονήθηκε από την ομάδα Γεώπα της ΚΟΠΑ, που είναι η ομάδα των εργοδοτών, που μέλη της ε, είναι εθνικές γεωργικές οργανώσεις, που είναι είτε μέλη της ΚΟΠΑ, είτε εγκεκριμένοι από την ΚΟΠΑ να γίνουν μέλη της ΖΕΟΠΑ ΚΟΠΑ. Και έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικές συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο. Θα μας τα εξηγήσει λεπτομεριακά στην ακρόαση του κύριο Πότερμαν. Η Ζωπά Κοπά δημοσίευσε ε, έκθεση το Δεκέμβριο του 2014. Γενικώ ε, εκδίδει γνωμοδοτήσει επί προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανονισμού και οδηγίε που διαπούν την κοινωνική πολιτική και τον Δεκέμβριο του 2016 ε, εξέδωσαν έκθεση για τον κοινωνικό διάλογο, ζητώντας ε, περισσότερο και πιο διευρυμένο κοινωνικό διάλογο και απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η αδήλωτη εργασία. Θα πρέπει να βρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να βελτιωθεί η κατάσταση των εργαζομένων στο γεωργικό τομέα και να απλουστευτεί η γραφειοκρατία για τους εργοδότες. Το βασικό πρόβλημα του συστήματος είναι ότι η αδήλωτη και παράνομη εργασία προωθούν την κοινωνική απάτη και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων σχετικά με την πρόσληψη, την απασχόληση, τους φόρους και την κοινωνική ασφάλεια έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αυτό θα αποβεί προ όφελο των εργαζομένων, των γεωργών, των εργοδοτών, αλλά και των κρατών μελών. Και φυσικά κυρίως για όλους τους απασχολούμενους στη γεωργία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κρίς Πότερμαν, που είναι πρόεδρος της ΖΕΟΠΑ ΚΟΠΑ για 10 με 15 λεπτά, προκειμένου να μας παρουσιάσει την έκθεση και θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους ευρωβουλευτές. Έχετε το λόγο κύριε Πότερμον, κύριε Πρόεδρε της ΖΟΠΑΚΟΠΑ. Περιμένουμε την παρουσίαση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, την Επιτροπή σας και τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την έκθεση που εκπονήσαμε μαζί με τα μέλη της ΖΕΟΠΑ. Είναι μια σύντομη παρουσίαση των πεπραγμένων μας και των αποτελεσμάτων και των πορισμάτων. Εισαγωγικά ο πρόεδρος Σικέσκης σας είπε τι είναι η ΤΖΕΟΠΑ. Ξέρετε ότι είμαστε η ομάδα των εργοδοτών που συνεργαζόμαστε με την ΚΟΠΑ και όπως είπε ε, στην εισαγωγή του ο Πρόεδρος μπορούμε να έχουμε με τα συνδικάτα διάλογο, κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη και ε, συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος ε, μίλησε ήδη εισαγωγικά για την οργάνωσή μας. Είχαμε την ευκαιρία στα τέλη του 2014 να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και με χαρά Αναλάβαμε αυτή τη μελέτη, το σεμινάριο ουσιαστικά για την αδήλωτη παράνομη εργασία στη Γεωργία ανά την Ευρώπη. Για ποιο λόγο θελήσαμε να διοργανώσουμε και να εκπονήσουμε μια τέτοια μελέτη. Η αδήλωτη εργασία οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ και το ίδιο το κοινωνικό ντάμπινγκ σε αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε γιατί είναι εις βάρος των Ε, εργοδοτών οι οποίοι ε, τηρούν τους νόμους και τους κανόνες. Θα πρέπει να παταχθεί η αδήλωτη εργασία, το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ε, τέσσερα είναι τα βήματα που ακολουθήσαμε. Σύντομα θα σας τα παρουσιάσω. Πρώτον, να δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και οι ορισμοί, αν υπάρχουν ορισμοί για το τι εστία αδήλωτη ή ε, παράνομη εργασία ή που υποδηλώνεται δεν στο σύνολό της. Το δεύτερο είναι σύστημα ελέγχου, πώς εργα... οργανώνεται ο κοινωνικός έλεγχος. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι το τρίτο, οι καλές πρακτικές, οι βέλτιστες πρακτικές και στο τέταρτο στάδιο προχωρούμε σε συστάσεις και συμπεράσματα. Στην αρχή της παρουσίασης θέλω να πω ότι η μελέτη που κάναμε διατίθεται σε έξι γλώσσες, έξι γλώσσες αν θέλετε μπορείτε να τη λάβετε σε μία από τις γλώσσες της αρεσκίας σας. Και βεβαίως ε, υπάρχει και σημερινή παρουσίαση PowerPoint, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα να σας τη δώσουμε. Καταρχάς να πω μερικά λόγια για τους ορισμούς, πολύ σύντομα. Όταν κάνουμε την εξής ερώτηση, πώς μπορούμε να ορίσουμε την αδήλωτη εργασία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομικά δεσμευτικός ορισμός της εργασία, εργασίας, μαύρης εργασίας ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα έγγραφο του 1998 και ένα άλλο του 2007 όπου αναφέρεται ότι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει ε, αυτό τον όρο αδείλωτη εργασία. Είναι οποιαδήποτε αμοιβόμενη νόμιμη εργασία η οποία δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές. Αυτό είναι ορισμός από τα έγγραφα του 1998 και του 2007. Όταν μιλούμε για δήλωτη εργασία δεν δηλώνεται στις κρατικές αρχές αλλά καλύπτει φάσμα δραστηριοτήτων, ε, υπηρεσίες, οικιακή βοηθός, παράνομη εργασία, εργασία ε, ανθρώπων χωρίς χαρτιά κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν πανευρωπαϊκή ε, ρύθμιση ή δεσμευτικός ορισμός. Η παράνομη εργασία τι είναι. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει οδηγία του 2009 για παράνομα διαμένονται στην Ευρώπη πολίτες τρίτων χωρών που εργάζονται και στο άρθρο 2 γίνεται λόγος για απασχόληση Ενό ε, πολίτη τρίτη χώρα που διαμένει παράνομα. Έτσι ορίζεται η παράνομη εργασία. Τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν και δήλωσαν ότι σε 18 ε, κράτη-μέλη η παράνομη εργασία είναι από μόνη της ε, ποινικά κολάσιμη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν ορισμοί. Σε κάποιες χώρες όμως η αδήλωτη εργασία είναι ένα είδο παράνομη εργασία. Στη Γαλλία, Πορτογαλία, Γερμανία και σε άλλες χώρες. Όπως βλέπετε από τη διαφάνεια, η παράνομη εργασία είναι τελείως διαφορετική από την αδήλωτη. Και σε κάποιες άλλες επικρατεί σύγχυση δεν υπάρχει καμία μορφή ορισμού. Για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Αν θέλει κάποιο να κάνει κάτι κατά τη αδήλωτη εργασία και τη παράνομη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε του ίδιου ορισμού σε όλη την Ευρώπη για να καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα στο τέλο. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε όταν γίνεται λόγος για κοινωνικό dumping είναι οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι και αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αδήλωτη εργασία. Δεν υπάρχει ορισμός εδώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αν κοιτάξουμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα διαπιστώσουμε και στη σελίδα 19 της μελέτης αναφέρουμε διάφορες περιπτώσεις, ε, υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχει ένα είδος ορισμού. Οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι ποιοι είναι. Είναι κάποιοι που προσλαμβάνονται ε, με το στην εθνική νομοθεσία ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά πάντα εργάζονται ως υπάλληλοι. Δεν ε, ε, έχουν ελευθερία να αποφασίζουν το χρόνο, το περιεχόμενο, ούτε τον τόπο εργασίας, ούτε συμμερίζονται τον επιχειρηματικό εμπορικό κίνδυνο του εργοδότη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας υπάλληλος που προβάλλεται ή δηλώνεται ως αυτοαποσχολούμενος. Και ένα τελευταίο στοιχείο από τους ορισμούς. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε συζήτηση με τα μέλη μας και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, εκείνους που ασχολούνται με την απόσπαση εργαζομένων. Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει απόσπαση εργαζομένων στη Γεωργία. Δεν ισχύει αυτό. υπάρχουν επίσης χώρε όπω είναι η Γαλλία, όπου αυξάνεται η απόσπαση εργαζομένων. Ε, κυρίως αυτοί εργάζονται στις οικοδομές, ε, στις μεταφορές και όχι στη γεωργία οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Ε, και ένα τελευταίο στοιχείο, όταν γίνεται λόγος για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, είναι πολύ δύσκολο και πάλι να βρούμε ορισμούς. Βλέπετε, εδώ είναι περισσότερο το κόκκινο το όχι παρά το ναι για τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Ε, επόμενο βήμα, ο έλεγχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, στο δεύτερο στάδιο συζητήσαμε πώς γίνεται η επιβολή των κανονισμών και των νόμων και τι γίνεται με την επιθεώρηση εργασίας. Ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Επίσης ε, ασχοληθήκαμε και με τις κυρώσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και Ποιο έχει την αστική ευθύνη. Έστειλαμε στα μέλη μας ε, κάποια ερωτηματολόγια και μία από τις ερωτήσεις που τους ε, θέσαμε ήταν να μάθουμε ποια είναι η νομοθεσία που διέπει την επιθεώρηση εργασίας. δεύτερο, τι δικαιώματα και τι εξουσίες έχουν οι εργασίας και τι δικαιώματα ε, έχουν οι εταιρείες ε, οι επιχειρήσεις στις οποίες γίνονται επιθεωρήσεις. Και στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ε, ουσιαστικά ασχολείται με την επιβολή του νόμου. Και υπάρχουν συστήματα που βασίζονται στην ε, αποτροπή και αλλού συστήματα που βασίζονται στη συμμόρφωση. Η περισσότερη πρόληψη είναι πολύ σημαντική βέβαια, και είχαμε την ευκαιρία να ε, μελετήσουμε και το εξή. Έχουμε παραδείγματα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες μέλη όπου υπάρχουν και άλλα μέσα ε, Συλλογικέ συμβάσεις, νομοθεσία εκτός από την επιθεώρηση εργασίας ή απλούστευση της διοίκησης. Θα το δούμε στη συνέχεια, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη πάνω από 20 εκατομμύρια είναι οι εργαζόμενοι στη γεωργία, αλλά από χώρα σε χώρα είναι πολλέ διαφορέ. Σε χώρε όπω είναι η Γερμανία, η Σουηδία, έχουμε εργαζομένου πλήρους απασχόλησης που εργάζονται στις εταιρείες, σε εκμεταλλευσει όλο το χρόνο. Σε άλλε χώρε όπω είναι η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, έχουμε εποχιακού εργαζομένου και συμβάσει πολύ μικρού χρόνου μηνών. Η οργάνωση εργασία είναι πολύ διαφορετική. Και ένα τελευταίο, σε πολλές χώρες ε, βλέπουμε να έχουμε όλο και περισσότερο ε, έναν εργαζόμενο που έχει μία σύμβαση αλλά εργάζεται για πολλούς εργοδότες ταυτόχρονα. Είναι συνεργοδότηση ας πούμε. Προχωρώ στην απλούστευση. Να σας δώσω δύο σύντομα παραδείγματα. Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεκριμένη διαφάνεια Ποια είναι η επίσημη δήλωση που πρέπει να κάνει ε, ο εργοδότης. Ποια στιγμή πρέπει να δηλώσει ε, τη σύμβαση. Όταν αρχίζει να ισχύει, ε, πριν αρχίζει να ισχύει η σύμβαση ή μετά. Γερμανία, Πολωνία, Πορτογαλία. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα γίνει αυτή η κοινοποίηση ή η δήλωση. Μπορεί να είναι έγγραφη ή μπορεί να είναι ηλεκτρονική. Και ένα τελευταίο Πόσες φορές πρέπει να γίνει αυτή η δήλωση άπαξ ή πολλές φορές. Αν χρειαστεί κάποιο να το δηλώνει μία και μόνη φορά, είναι πιο εύκολο. Μπορεί κανεί να είναι νομοταγή. Όταν είναι περίπλοκη η διαδικασία, ε, έχουμε και σφάλματα και προβλήματα. Αυτή η διαφάνεια τώρα εδώ που σα δείχνω είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη δήλωση που έχει κάνει ο εργοδότης, μπορεί να υπάρχουν λάθη, για να μην είναι 100% λάνθαστε. Όταν υπάρχει έστω και το παραμικρό σφάλμα, τι γίνεται και ρωτήσαμε. Σε πολλές χώρες, ακόμα και ένα τυπικό σφάλμα, θεωρείται αδήλωτη εργασία και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο στις χώρες με πράσινο είναι διαφορετική αντιμετώπιση επάνω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και οι κυρώσεις ποιες θα είναι, να είναι με την ε, τασταλία. Ε, δηλαδή, άλλο είναι να έχεις κάνει ένα λάθος στη δήλωση, τυπικό, και ε, ναι, δεν μπορεί να θεωρείται αδήλωτη εργασία εξορισμού αυτό. Για τις διαδικασίες τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης όταν κάποιος εργάζεται στην εκμετάλλευσή του και ποια είναι η σχέση εργασίας. Υπάρχουν πολλές διοικητικές υποχρεώσεις, και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αν, αν δείτε από κάτω όμως τι γίνεται με την κοινωνική ασφάλιση και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι πολλά τα έγγραφα. Και υπάρχει μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή για τη Γεωργία και παρακαλώ την προσοχή σας. Άλλαξαν οι, αγώνες, ε, κανόνες συγγνώμη, για την εποχική εργασία και πολλοί εργαζόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη επασχολούνται στη Δυτική Ευρώπη και κάθε εργοδότης θα πρέπει να δηλώνει ε, την εργασία ε, και το μισθό ε, στη χώρα καταγωγής του εποχιακού εργαζομένου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους εργοδότες. Ένα τελευταίο στοιχείο και μετά θα προχωρήσω πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σε οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Είδαμε στις χώρες αυτές που συμμετέχουν και είναι πάρα πολύ ισχυρές οι οργανώσεις των εργοδοτών βοηθούν ε, τους εργοδότες να συμμορφώνονται με τον κανόνα. Εδώ βλέπουμε πώς οργανώνεται ο κοινωνικός διάλογος. Το επόμενο δεν θα το σχολιάσω στη διαφάνεια. Μπορείτε να το δείτε στην έκθεση, είναι γύρω στις 15 σελίδες. Ψάξαμε τις καλές πρακτικές στις χώρες μας και έχουμε καλές πρακτικές και για την ομοθεσία και για να δούμε τι γίνεται με την επιθεώρηση εργασίας και πώς συνεργάζονται οι εργοδότες σε διάφορες χώρες με παραδείγματα. Έχουμε καλές πρακτικές επίσης στην επιβολή του νόμου, στην απλούστευση. Και τέλος, πώς οργανώνεται ο κοινωνικός διάλογος εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο και για τη δική σας δουλειά. Σας είπα ότι υπάρχει σε έξι γλώσσες η μελέτη μας. Μπορείτε να προμηθευτείτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει. Και στο τέλος έχουμε ένα κεφάλαιο μόνο με συμπεράσματα και συστάσεις. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποια. Έχουμε κάποιες συστάσεις για τους ορισμούς. Όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινό ορισμός. Κοιτάξτε στις συστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε γνώση των εθνικών ορισμών και κάτι να γίνει στο μέλλον. Δεύτερον, στοιχείο, στα συμπεράσματα. Τι μπορεί να κάνει μια χώρα. Και στις συστάσεις το λέμε. Χρειάζονται μέτρα προληπτικά. Τρίτο στοιχείο. Να είναι αναλογικές οι κυρώσεις. Δεν μπορεί να έχει κάνει ένα τυπικό σφάλμα και να θεωρείται αδήλωτη εργασία ή να έχει την ίδια αντιμετώπιση στις κυρώσεις. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η να εχει την ιδια αντιμετωπιση στις κυρωσεις πολυ σημαντικο θα μεινει η απλουστευση των διαδικασιών και των ε, γραφειοκρατικών, γιατί όσο βαρύτερη η διαδικασία, τόσο μειώνεται η συμμόρφωση. Οι καλές πρακτικές βοηθούν και στη γεωργία έχουμε πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Δεν έχουν, ας πούμε, έναν εργαζόμενο στο γραφείο για να ασχολείται με όλο αυτό το διοικητικό σκέλος. Επίσης υπάρχουν τα συστήματα συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και την επιθεώρηση εργασίας, αυτή η τριμερής ε, συνεργασία και είναι σημαντικό ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Στις χώρες, όπως είπα, όπου υπάρχουν ισχυρές οργανώσεις, ε, οργανωμένες, οι ε, κανόνες εφαρμόζονται καλύτερα. Ένα τελευταίο. Η παράνομη και αδήλωτη εργασία δεν είναι μόνο το πρόβλημα, πρόβλημα μάλλον για την συγκεκριμένη χώρα είναι και διεθνές. Εμείς είμαστε παρατηρητές στην πλατφόρμα ε, για την αδήλωτη εργασία και την επόμενη διετία θα ασχοληθούμε και με τη γεωργία εκεί και θα υποβάλουμε τις συστάσεις μας για καλές πρακτικές και απλοποίηση για benchmarking, συγκριτική αξιολόγηση κτλ. Συμπέρασμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη. Εμείς είμαστε κατά κάθε είδους κοινωνικής ε, ε, απάτης, απάτης στην εργασία και αδήλωτης εργασίας Αλλά αυτό που χρειάζονται οι χώρες και η Ευρώπη δεν είναι περισσότερη νομοθεσία, αλλά καλύτερη νομοθεσία και απλούς κανόνες για να εφαρμόζονται από τα μέλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που τηρήσατε το χρόνο σας. Θα περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτο ζήτησε το λόγο ο κύριος Λουαζό. Παρακαλώ κύριε Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το περασμένο Φεβρουάριο σε μια αποστολή στην Γαλλία με τον κύριο Φεράν συνάντησα ε, αγρότες από το Βοκλούς και μας είπαν και μερικά αξιοπερίεργα πράγματα. Είπαν ότι χιλιάδες αποσπασμένοι εργαζόμενοι εργάζονταν στον τομέα αυτό, στο, στο διαμέρισμα Βοκλούς. Χρειάζεται πολύ, πολλά εργατικά χέρια γιατί δεν είναι μηχανοποιημένος ο κλάδος. Επίσης, ε, υπάρχει ε, συμφωνία με την Ισπανία ε, και γίνεται εισαγωγή εργαζομένων και από τη Λατινική Αμερική. Στο Βοκλούζ έχουμε ε, Περουβιανούς, ε, Χιλιανούς με εξάμηνες συμβάσεις για την συλλογή των αποδοκιπευτικών. Τι πρέπει να κάνουμε για την προέλευση των εργαζομένων. Θα πρέπει να είναι Ευρωπαίοι και επίσης να αναβαθμίσουμε και να εξάρουμε το γεωργικό τη γεωργική εργασία και γίνει και άνισο και το κόστος της εργασίας. Βέβαια, κάθε κράτος θα πρέπει να ελέγχει τα σύνορά του και να έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει την αγορά εργασίας του. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπότερμαν, τον πρόεδρο της ε, ΧΕΟΠΑ, τον είχα συναντήσει για μια προκατακτική παρουσίαση της έκθεσης και χαίρομαι για τη συζήτηση που έχουμε εδώ, γιατί πολλά λέμε για τη γεωργία και για τους επαγγελματίες στη γεωργία, αλλά άλλο η γεωργική απασχόληση ε, που δεν, πρέπει, που δεν είναι να μελούμε και να μην ξεχνούμε και τους ε, εργοδότες ε, στο γεωργικό κλάδο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις αδικίες και το κοινωνικό ντάμπινγκ και στη γεωργική απασχόληση. Είμαστε υπέρ τη αηφορία φυσικά στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να είμαστε υπέρ και τη κοινωνική αηφορία. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση και χαίρομαι που την εκπονήσατε και εμείς τη συζητούμε. Θα μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών θεμάτων. Είπατε ότι δεν θέλουμε περισσότερη νομοθετική ρυθμίση, αλλά βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και αν σας κατάλαβα καλά, ήδη υπάρχει μια πρόταση για την εναρμόνιση των ενιών και των ορισμών. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί και έννοια στα κράτη-μέλη. Οπότε, εξ ε, των πραγμάτων δημιουργείται άνηση μεταχείριση από χώρα σε χώρα. Και επίσης όχι μόνο άνηση μεταχείριση υπάρχει, αλλά και διαφορετικές κυρώσεις. Οπότε είναι κατάφορη η διαφορά στην αντιμετώπιση της αδήλωτης ή παράνομης εργασίας. Αυτό που ζητήσατε, αυτό που κατάλαβα τουλάχιστον, είναι να γίνει εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας, για να υπάρχουν ομοιόμορφοι ορισμοί. Ε, και μια άλλη διευκρίνηση θα ήθελα να ζητήσω. Η γεωρική διεργασία ε, είναι αβέβαιη, εξαρτάται από, πολλές, ε, από πολλούς αστάθμιτους παράγοντες και πολλές φορές απαιτεί μέσα σε ένα μήνα, σε 40-45 μέρες, ε, πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό και μια μεγάλη συγκέντρωση και ένα εργατικό δυναμικό που θα πρέπει να μπορεί να κινείται από τη μία απασχόληση στην άλλη με μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί εποχιακά εργαζόμενοι και εδώ και 20, 30, 40 χρόνια όταν ξεκίνησε η μετανάστευση από την Ισπανία στην Γαλλία μόνο για τον τρίγο με ε, βραχυπρόθεσμες συμβάσει και συνεχίζεται τέτοια αποδημία μόνο και μόνο για την εποχιακή εργασία του ε, τρίγου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αποφύγουμε αυτή η εντατικοποίηση σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα να μην ενισχύσει το φαινόμενο του κοινωνικού τάμπη και της ανισότητας. Γιατί η γεωργία θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, να λαμβάνει όμως υπόψη και το μισθολογικό κόστος, το εργασιακό κόστος. Επίσης και η ρυθμίση των μισθών ε, συνήθως διαθετείται από συλλογικές συμβάσεις και μερικές φορές είναι και περιφερειακού χαρακτήρα, τουλάχιστον στην Ισπανία. Οπότε υπάρχουν ε, διαφορές ακόμη και εντός της ίδιας χώρας μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ε, για τον υπολογισμό του κόστου αυτή τη ε, συλλογική ρύθμιση. Υπάρχει κάποιο τρόπο με τον οποίο εμεί θα μπορούσαμε να παρεύουμε, κύριε Μπότερμαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δενανό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση, γιατί έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Γεωργία, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η Γεωργία εδώ. Και όντω δεν υπάρχει νέος ορισμό για την παράνομη εργασία, για την αδήλωτη εργασία. Οπότε, τι κάνει η Ευρώπη για όλα αυτά τα θέματα, αν δεν έχει καταφέρει να θεσπίσει κάποιου ενιαίου ορισμού. Και πραγματικά ο κίνδυνο θα είναι να μείνουμε τα χέρια σταυρωμένα, γιατί θα οδηγηθούμε σε στρέβλωση ανταγωνισμού. Ήδη διαπιστώσατε αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ε, κάποιο αδήλωτο ε, είναι σαν να είναι ανύπαρκτο, αόρατο, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα κοινωνική ασφάλιση ή ε, υγειονομική περίθαλψη. Οπότε υπάρχει και ουσιαστικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να αγγίψουμε σε αυτό το θέμα. Με έχει απασχολήσει γιατί ιδιαίτερα για την συγκομιδή μήλων έχουμε έντονα εποχιακό χαρακτήρα και στην δική μου γενέτειρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε μία σύμβαση που να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες εποχές ώστε να συνδυάζονται αυτές οι εποχιακές εργασίες για να καταλήξουμε σε ε, μόνιμες συμβάσεις. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη χαρά την παρουσίαση της έκθεσης ε, της ΓΕΟΠΑΚΟΠΑ ε, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι οξύ και θα πρέπει να αναζητήσουμε ευέλικτες λύσεις ώστε να μην είναι η θεραπεία χειρότερη από την ασθένεια. Ε, στις ε, γεωργικές περιοχές ή στην υπεθρό αγροτικές ζώνες ε, ο κόσμος εγκαταλείπει τις εργασίες του και μετακομίζει στις μεγαλύτερες πόλεις. Οπότε, αν ενισχυθούν οι διατυπώσεις, θα οξυνθεί αυτό το φαινόμενο της αστιφιλίας ή της απερίμωσης της υπαίθρου. Στην έκθεσή σας επίσης ε, απαριθμίσατε τους, κατα... λόγους για τους οποίους έχουμε παράνομη αδήλωτη εργασία. Ίσως ε, σε κάποιες χώρες ε, τα φορολογικά συστήματα είναι δυσβάσταχτα και αποτρέπουν τους εργοδότες από το να δηλώσουν τους απασχολούμενους τους. Ή υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία, πολλές διοικητικές διατυπώσεις και γι' αυτό οι εργοδότες μερικές φορές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να μην δηλώσουν τους εργαζομένους τους. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε ευέλικτους τρόπους και να δώσουμε κίνητρα στους εργοδότες για να δηλώνουν τους απασχολουμένους τους. Γιατί σήμερα η κατάσταση μπορεί να μην τους ευνοεί, αλλά στο μέλλον μια τέτοια προτροπή ε, θα μπορούσε να ήταν και ευνοϊκή. Και τα κίνητρα δεν ε, θα πρέπει να είναι κατά ανάγκη οικονομικά, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους εργοδότες για να δηλώνουν ε, τους ε, εργαζομένους τους ώστε να μπει μια τάξη σε αυτό το σύστημα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μας είπατε όμως ποιο είναι το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας στη Γεωργία. Είναι 1%, 50%. Να έχουμε μια ε, αίσθηση της τάξης μεγέθους. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, περίοδοι ε, με έντονη γεωργική απασχόληση, αλλά άλλες εποχές δεν χρειάζονται ιδιαίτερα εργατικό δυναμικό στη γεωργία. Επίσης, η ορολογία είναι σημαντική. Εξισώσατε την αδήλωτη εργασία με το κοινωνικό ντάμπικ. Σε, άλλες, σε άλλους τομείς όμως, όπως τις μεταφορές, αναφέρονται ότι και οι, δια, οι μισθολογικές διαφορές μερικές φορές συνιστούν κοινωνικό ντάμπινγκ. Οπότε τι ισχύει τελικά. Είναι κοινωνικό ντάμπινγκ αν πληρώνω εγώ τον εργαζόμενο μου κάτω από 2.000 ευρώ. Ή είναι κοινωνικό ντάμπινγκ όταν δεν το δηλώνω. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ακριβείς διατάξεις. Άλλο αδήλωτη εργασία και άλλο το ύψος των μισθών ή το ύψος της αμοιβή που καταβάλλεται για τη συγκεκριμένη εργασία. Δεν θα πρέπει για διαφορετικά πράγματα να χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη ορολογία. Επίσης, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φροντίσουμε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών. Ευχαριστώ κύριο Σκαπούτο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μπότερμαν για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση η οποία βοηθά το διάλογο μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και γεωργών. Ένα διάλογο τον οποίο θα πρέπει να ε, παρακολουθούμε και να φροντίζουμε όλοι. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο για το θέμα αυτό, ιδιαίτερα για την ε, αδήλωτη εργασία, γιατί προέρχομαι από την περιοχή της Καμπανίας στην Ιταλία, όπου η πτυχή αυτή έχει προσλάβει και διαστάσεις κατεπήγοντος στην πραγματικότητα. Ε, είναι μία μορφή υπόγειας μαύρης εργασίας που είναι η πιο ε, ανησυχητική στον γεωργικό τομέα όταν υπάρχει ένας διαμεσολαβητής ο οποίος δεν έχει καμία εξουσιοδότηση φυσικά ε, και καταχράται με εγκληματικό τρόπο ε, κάποιες ε, δομές για να εκμεταλλευτεί τον γεωργικό ε, στο γεωργικό τομέα κάποια κενά του συστήματος. Ε, στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη αντίδραση, ε, υπήρξε έγκριση συγκεκριμένης νομοθεσίας για αυτή την αδήλωτη εργασία και θεωρώ ότι είναι και μια βέλτιστη πρακτική την οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η ευθύνη είναι αυτού ο οποίος εκμεταλλεύεται τη μαύρη εργασία. Δεν βλέπω όμω ε, αντίστοιχη ευαισθητοποίηση στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Τον περασμένο Μάιο υπέβαλα προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της αδήλωτη εργασίας και ε, των μεσολαβητών αυτών και δεν ε, ικανοποιήθηκα από την απάντηση, γι' αυτό και υπέβαλα μια δεύτερη ε, προσπαθώντας να ε, διευκρινίσω και τις ιδιαιτερότητες και το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το φαινόμενο. Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου διαφεύγει στη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ότι ε, η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εργασιακή ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση δεν επιλύουν το πρόβλημα, διότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πέφτουν στα δίχτυα αυτού του δικτύου είναι αόρατοι για το σύστημα θα πρέπει στην πραγματικότητα να ληφθούν ε, μία σειρά από μέτρα τα οποία θα επιτρέπουν μεγαλύτερες παρεμβάσεις του κράτους, ξεκινώντας για παράδειγμα από κάποια εργαλεία ε, τα οποία θα θέτουν και όρους στην κοινή γεωργική πολιτική και θα υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις ε, για τη δημιουργία κατάλληλων δομών που θα δημιουργηθούν με κατάλληλο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς. Η ουσιαστική ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι η εξής. Θεωρείτε ότι αν υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία των θεσμικών οργάνων και του δημοσίου τομέα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την επίλυση αυτού του προβλήματος, που είναι και ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία πλήττουν το γεωργικό τομέα. Κυρία όχι, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση. Διάβασα την επικεφαλίδα και έχει σημασία για μένα αυτό. Είναι σημαντικό ως Επιτροπή Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατρανώσουμε ότι οποιαδήποτε αδήλωτη εργασία, παράνομη εργασία, μαύρη εργασία ε, και προσπάθεια ατασταλίας ε, το καταδικάζουμε στεναρά δεν είναι πτέσμα. Δυστυχώς σε πολλά κράτη, σε πολλά μέρη θεωρείται πτέσμα, ένα ε, μικρό παράπτωμα. Καθόλου. Θα πρέπει να το πούμε και να το λένε. Δεν το είπαν οι προλαλήσαντες, να είναι σωστές οι κυρώσεις και πραγματικά όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους, δεν τους δηλώνουν και πολλές φορές είναι πρόσφυγοι και μετανάστες και τους εργοδοτούν διότι είναι φθηνοί, θα πρέπει να διώκονται και ποινικά. Δεν είναι πτέσμα, επαναλαμβάνω. Και θα πρέπει να βρούμε πιο σταρά τα λόγια για να τα πούμε όλα αυτά. Και τα γνωρίζουν πολύ συχνά οι αγρότες, οι εστιατορές, ότι ο γείτονα ε, απασχολεί παράνομους. Ε, αν δεν το ξέρουν, το υποπτεύονται, το θεωρούν ε, ότι καλά δεν τρέχει και τίποτα, αλλιώ η εταιρεία δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και θα έκλεινε. Όχι. Ε, η παράνομη εργασία, η παράνομη απασχόληση είναι κάτι το οποίο καταδικάζουμε απερίφραστα. Και δεν μπορούμε να βρίσκουμε δικαιολογίε για τη φορολογία, για τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν έχει σημασία. Όποιο δεν απασχολεί ανθρώπου με σωστό τρόπο, ε, ε, κάνει κάτι το οποίο είναι ποινικά κολάσιμο. Και στη Βαβαρία το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι μόνο στην οικοδομή και στη γεωργία. Και είναι πραγματικά επονίδιστο αυτό για μια χώρα σαν τη Γερμανία και ένα κρατήδε σαν τη Βαβάρια. Να τα λέμε έξω από το δόν για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Καλωσορίζω και εγώ τους καλεσμένους μας. Ε, τον ευχαριστώ θερμά για την πολύ αξιοθαύμαστη αυτή έκθεση ε, που όμως χρησιμοποιεί δεδομένα από 16 χώρες μέλη. Πότε επιτέλους ε, μπορούμε να περιμένουμε συμπερίληψη και της Κροατίας στις χώρες από τις οποίες συγκεντρώνεται στοιχεία. Αναφέρατε και τρία παραδείγματα καλών πρακτικών που ίσως για μερικές χώρες είναι υπερβολικά φιλόδοξα. Γιατί δυστυχώς δεν είναι παντού οργανωμένοι οι γεωργοί σε συνδικάτα ή σε οργανώσεις ή συνεταιρισμούς για να έχουν διαπραγματευτική ισχύ ε, στις συζητήση με τους κοινωνικούς διαλόγους και σίγουρα κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό και θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση μια τέτοια μεγάλη, μεγάλη οργάνωση αλλά δυστυχώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι δεν καταφέρουν καν να συμφωνήσουν στην οδηγία για το ωράριο εργασία. Πολλό δε μάλλον στη Γεωργία που δεν είναι καλά οργανωμένη η Γεωργοί παντού ώστε να μπορούν με πυγμή να δίνουν μάχη για τα δικαιώματά τους. Επίσης είπατε ότι το πρόβλημα των χωρών μελών δεν είναι η έλλειψη κανονιστικών διατάξεων, αλλά οι κακές κανονιστικές διατάξεις. Ε, μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα τι πιστεύετε θα μπορούσαν να κάνουν οι νομοθέτες, πώς να βελτιώσουμε την νομοθεσία για να βελτιώσουμε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της Γεωργίας. Όταν ε, εισηγήτρια της έκθεσης για το ρόλο των γυναικών στην Ήπεθρο, είχαμε μία ακρόαση στην οποία μιλήσαμε για την αναγνώριση ε, του καθεστώτος ε, των ε, συζύγων γεωργών ε, και τις θέσεις τους στην γεωργική εκμετάλλευση. Τα κράτη-μέλη ε, είναι έτοιμα να δεχτούν κάτι τέτοιο και να το συμπεριλάβουν στην νομοθεσία για να αναγνωρίσουν το ρόλο των γυναικών στην Ήπεθρο και την παρουσία τους ε, στην οικογενειακή εκμετάλλευση γιατί με την εργασία τους πραγματικά βοηθούν ε, στην άσκηση γεωρικών δραστηριοτήτων στην οικογενειακή εκμετάλλευση. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση θα έλεγα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι οι χιλιάδες πρόσφυγες και κυρίως οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν εισέλθει στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν πλέον εγκλωβιστεί είτε στην Ελλάδα είτε στην Ιταλία. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι βεβαίω να υπάρχει μια παράνομη, μια μαύρη εργασία στον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει μια κρίση για τους μικροκαλλιεργητές, διότι οι φτωχοί αγρότες βρίσκονται σήμερα κάτω από την πίεση της Τρόικας. Η Τρόικα έχει επιβάλει φορομπηκτικές πολιτικές, γίνονται κατασχέσεις αγροτικής γης, και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαδικασία όπου φτωχοποιούνται συνεχώς οι Έλληνες αγρότες και ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται σε αγροτικές εργασίες κυρίως για μεγαλοκαλλιεργητές. Με αποτέλεσμα στην ουσία να διαλύεται η μικρή οικογενειακή αγροτική επιχείρηση, οι μεγαλοκαλλιεργητές να αξιοποιούν παράνομα αυτή την εργασία και ταυτόχρονα πλέον να κερδίζουν και να λειτουργούν αθέμητα έναντι των φτωχών αγροτών. Το επόμενο στοιχείο που παρακολουθούμε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να δώσει σε δίθεν πρόσφυγες ταυτόχρονα κρατική γη να την καλλιεργήσουν. Δηλαδή την ώρα που αρπάζουν οι, εφορίε εφορίες και το δημόσιο κατάσχει την γη των Ελλήνων αγροτών, ταυτόχρονα θέλουν να δώσουν, έτσι δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Αποστόλου, τουλάχιστον σε 1.500 άτομα που τους αποκαλεί πρόσφυγες να τους δώσει γη να καλλιεργούν. Και το επόμενο στοιχείο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι θέλουν να ιδρύσουν τις επωνομαζόμενες ειδικέ οικονομικές ζώνες, όπου εκεί δεν θα ισχύει η εργατική νομοθεσία, θα μπορούν να δουλεύουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Πρόσφυγες έτσι λένε ότι είναι, αλλά μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι πρόσφυγες από την ώρα που κάνουν αίτηση μέχρι να πάρουν το καθεστώ πρόσφυγα περνάνε τρία ή τέσσερα χρόνια. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα δουλεύουν με εργασιακέ σχέσει οι οποίε δεν θα δεσμεύονται από την νομοθεσία, δεν θα υπάρχει κοινωνική ασφάλιση για αυτού και δεν θα υπάρχει το μήνυμα των αμοιβών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο για την Ελλάδα, φαντάζομαι και για την Ιταλία και την Ισπανία και θα πρέπει η έκθεση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Διότι έτσι καταστρέφονται πλέον οι φτωχοί Ευρωπαίοι αγρότες και αξιοποιούν οι μέγαλο αγρότες τους, ε, τα εκατομμύρια των παράνομων, παράνομων μεταναστών και τους βάζουν και δουλεύουν με συνθήκες μαύρης εργασίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, <clears throat> εξαντλήσαμε το κατάλογο των αγοριτών και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο για να euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τώρα σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μετέθησαν. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις ε, όπως τις σημείωσα εδώ στα σημειώσεις μου. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση για τους ε, πρόσφυγες. Ε, πολιτικοί πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται τώρα εδώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έγινε και μία μελέτη στα πλαίσια της ε, ΖΕΟΠΑ. Ζητήσαμε από τα μέλη μας να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ε, έχουμε εργαζομένους πρόσφυγες. Εδώ δεν πρόκειται για νόμιμη εργασία και φυσικά ε, κανείς ε, δεν είναι υπέρ της παράνομης εργασίας και της αδήλωτης εργασίας, επομένως προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, τιμωρήσουμε τέτοιες πρακτικές. Αλλά όταν έχουμε πολιτικές, πολιτικούς πρόσφυγες, ε, όλοι όσοι απάντησαν από τις διάφορες χώρες, ε, προσφέρεται η δυνατότητα, αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένη, να τους προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας ε, για 10-12 μήνες. Να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις λοιπόν σε κάποιε χώρε, οι οποίε δίνουν άδειε εργασίας για σύντομο περιορισμένο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κάποιους πολιτικούς πρόσφυγες. Ε, έχουμε λοιπόν απαντήσεις που μας έδωσαν τα μέλη μας ε, αυτού του τύπου. Τώρα, για την ερώτηση της κυρίας ε, Πετήρ. Έχουμε ερωτήσεις μόνο από 16 χώρες, απαντήσεις συγγνώμη μάλλον μόνο από 16 χώρες, αλλά ο στόχος μας είναι να συμπληρώσουμε τις εργασίες μας. Πρόκειται ε, για ένα θέμα, το θέμα της αδήλωτης εργασίας ε, που μας απασχολεί. Είμαστε και παρατηρητές ε, στο εργαστήριο κατά της αδήλωτης εργασίας και ελπίζουμε μέχρι το 2019 που θα συζητηθεί και η Γεωργία να μπορέσουμε να έχουμε συμπληρώσει τη μελέτη μας και να έχουμε και απαντήσεις και από την Κροατία αλλά και από άλλες χώρες οι οποίες προς το παρόν δεν περιλαμβάνονται ε, στην έκθεσή μας. Ρωτήσατε επίσης κάποια πράγματα για την ποιότητα της νομοθεσίας. Ε, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές χώρες έχουν ψηφιστεί νόμοι με καλές προθέσεις αλλά διαπιστώνουμε ότι οι κανόνε είναι πολύ περίπλοκοι, ε, διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι σε αρκετέ περιπτώσει υπάρχουν οικογενειακέ γεωργικέ εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των γεωργών δεν έχουν μόνιμη εργασία στη διάρκεια του έτου, ε, είναι εποχιακή απασχόληση μόνο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν λοιπόν ανθρώπινοι πόροι, πρέπει να κάνουν τα πάντα μόνοι του. Ε, υπάρχει νομοθεσία λοιπόν για τα φετεογειονομικά προϊόντα, για την κτηνοτροφία κλπ ε, όλα αυτά αφορούν όμως τον ίδιο εργοδότη. Για αυτές τις μικρές λοιπόν γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να έχουμε μια νομοθεσία, ίσως να παραμείνει και συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά να πλουστευτούν οι κανόνες, όπως σας έδειξα το παράδειγμα. Για παράδειγμα, όταν γίνεται μια δήλωση ε, για την έναρξη κάποιων εργασιακών σχέσεων μπορεί σε κάποια χώρα να απαιτούνται αρκετά έγγραφα. Εάν αυτό λοιπόν περιορίζεται σε μία απλοποιημένη δήλωση θα μπορούσαμε να ε, βελτιώσουμε και την ποιότητα. Ε, είπατε κι εσείς ότι σε κάποιες χώρες η γεωργία δεν είναι πάντα πολύ καλά οργανωμένοι Νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος της ΕΟΠΑ και στις προσπάθειες που κάνουμε, το κάνουμε και στην Πολωνία και στη Βουλγαρία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους στις νέες χώρες και να τους εξηγήσουμε ε, πόσο σημαντική είναι και η κοινωνική εταίρη και πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον κοινωνικό διάλογο. Να υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων λοιπόν που θα λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Ε, εάν το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να λάβουν αποφάσεις, πάντα θα λαμβάνονται σε γενικό επίπεδο χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πράξη και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σε κάποιες χώρες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ε, τελευταίο στοιχείο, αυτοί οι διαμεσολαβητές είναι οι σύζυγοι που βοηθούν, διαπιστώσαμε ότι σε πολλές χώρες οι σύζυγοι ε, είναι αυτές οι οποίες εργάζονται και στο χωράφι, αλλά είναι αόρατες, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς ε, και συζητήσαμε και με την οργάνωση γυναικών της ΚΟΠΑ. Σε κάποιες χώρες ε, ξεκινάμε λοιπόν να δίνουμε ένα συγκεκριμένο καθεστώς στις γυναίκες οι οποίες εργάζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά θα πρέπει ε, να λαμβάνουμε υπόψη ότι το κόστος είναι πιο σημαντικό φυσικά, αλλά θα πρέπει κάπως να προβάλλονται και αυτές οι γυναίκες, να γνωρίζουμε ποιες είναι. Ε, υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει, έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά ε, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Κάτι ακόμα το οποίο σημείωσα, είπατε ότι στη μελέτη δεν ανα... ή μάλλον να το πω αλλιώ. Είπατε τι είναι κοινωνικό dumping. Ε, σημαίνει να πληρώνουμε κάτω από τα 2.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ε, αν κάποιος είναι αδήλωτος, τι σημαίνει κοινωνικό dumping. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα πολύ απλό ορισμό. Έχουμε κοινωνικό dumping αν κάποιος εργάζεται σε μία χώρα και οι κανόνες που προβλέπονται στη χώρα αυτή σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή οι συμβάσεις οι οποίες ισχύουν, ε, τα ημερομίσθια, το κόστος ε, της εργασίας, ε, οι άδειες, οι αργίες δεν γίνονται σεβαστά. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, αν αναφερόμαστε στο κοινωνικό ντάμπινγκ, έχουμε πολύ κοινωνικό, αναφορά στο κοινωνικό ντάμπινγκ την περίπτωση απόσπασης. Μπορεί κάποιος να έρθει σε μια χώρα τη της Ευρώπης των 15 για παράδειγμα να εργαστεί, αλλά ξέρουμε ότι εκεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ίδια ε, πληρωμή, η ίδια αμοιβή ε, και πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες εργασίας στο χώρο εργασίας. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένας απλός ορισμός. Ο πρώτος ομιλητής είπε ότι ε, στη Γαλλία το κόστος ε, εργασίας δεν είναι το ίδιο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν ε, ορομήσεις, εργασίες, αμοιβές, ε, λαμβάνουμε υπόψη ε, τις ε, ώρες που εργάζεται κάποιος. υπάρχει νομοθεσία και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδότες και εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν και να έχουμε συλλογικές συμβάσεις στις οποίες θα καθορίζουμε και τα όρια. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχουν διαφορετικά όρια αναχώρα και αυτό είναι λογικό γιατί το κόστος ζωής δεν είναι το ίδιο στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά όταν υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει να λαμβάνεται και αυτή η υπόψη. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έρθει για παράδειγμα κάποιο ε, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στο Βέλγιο ή στην Ιταλία, θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνε ε, οι οποίοι ισχύουν στη χώρα στην οποία παρέχεται η εργασία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το δεχτούν όλοι. Ε, ρωτήσατε επίσης για τα ποσοστά της αδήλωτης και παράνομης εργασίας. Είναι δύσκολο αυτό να το γνωρίζουμε, γιατί αν κάποιος δεν δηλώνεται, αν έχουμε παράνομη εργασία, Στη σελίδα 12 της μελέτης μας έχουμε κάποιες μελέτες οι οποίες κάνουν κάποιες εκτιμήσεις για τα ποσοστά και τους αριθμούς. Ε, στις μελέτες αυτές λέγεται ότι δεν είναι εύκολο να το προσδιορίσουμε. Υπάρχει επίσης και το Συνδικάτο της Γεωργίας, το ΕΦΑΤ, το οποίο εκπώνησε μία μελέτη και λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ποσοστά. Μελέτησαν ε, όμως ε, την κατάσταση σε 9 ή 10 χώρες, θα το είδατε ίσως αυτό το έγγραφο της ΕΦΑΤ και αναφέρονται σε ένα ποσοστό το οποίο θεωρώ όμως ότι είναι λίγο υπερβολικό της τάξης του 20% και κάτι παραπάνω. Λένε όμως ότι αυτό είναι προβολή από στοιχεία που έχουν σε κάποιες χώρες και ότι είναι αδύνατο να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Ε, Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σίγουρα δηλωτή εργασία βεβαίω. δεν θα είχαμε κάνει την ε, μελέτη δάλος, αλλά ε, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή ποσοστά. Τώρα, ε, για την απάντηση στην ερώτηση γιατί υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ, γιατί υπάρχει αδήλωτη και παράνομη εργασία, νομίζω ότι υπάρχει μια έμεση απάντηση παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει άμεση, διότι θεωρώ ότι σε πολλές χώρες δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της πραγματικά παράνομης εργασίας και της πραγματικά δηλώτης εργασίας και από την άλλη το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές κάποιες τυπικές διαδικασίες. Ε, για παράδειγμα, αν πρόκειται απλώ για μια τυπική διαδικασία η οποία δεν γίνεται σεβαστή, σε κάθε χώρα αυτό θεωρείται ε, σαν αδήλωτη εργασία. Αυτό πάλι δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να γίνεται και κατάλληλη διάκριση μεταξύ αυτών. Ε, υπήρξαν κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Ο Γάλλος βουλευτή που μίλησε πρώτος είπε ότι σε κάποιες ε, χώρες, κυρίως στη Γαλλία, υπάρχουν ε, μετανάστες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική ε, και εργάζονται. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη των 28 έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και ε, ελεύθερη ε, κυκλοφορία εργατικού δυναμικού. Αυτή είναι η Ευρώπη των 28. Τώρα, αν κάποιος ο οποίος ζει σε άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εξαρτάται εκεί από κάθε χώρα. Η χώρα αποφασίζει ποιος μπορεί να εισέρχεται στη χώρα της. Ε, στη ΖΕΟΠΑ, για παράδειγμα, έχουμε συναδέλφους από τη Φιλανδία και εκεί υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία για να υπάρχει δυνατότητα ε, πρόσληψης εργαζομένων από τη Ρωσία. Η Πολωνία έχει συμφωνία με την Ουκρανία. Επομένως υπάρχει δυνατότητα να προσλαμβάνονται άτομα από την Ουκρανία στην Πολωνία. Ε, οι χώρες του Νότου ε, έχουν συμφωνίες με χώρες της ε, Βόρειας Αφρικής, κάποιες χώρες του Νότου, για να δυνα... τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν άτομα από εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από την κάθε χώρα, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες ε, οι οποίοι να προβλέπουν ποιος μπορεί να έρχεται και ποιος όχι. Αν έρχονται λοιπόν άτομα από τη Λατινική Αμερική σε κάποιες χώρες, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν κανόνες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, για τι ερωτήσεις της κυρίας ακυλέρα. Ρωτήσατε αν είμαστε υπέρ της εναρμόνισης σε κάποιους ορισμούς. Να πω ότι όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις διάφορες πλατφόρμες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι ορισμοί ισχύουν σε κάθε χώρα, να προσπαθήσουμε αν θέλουμε όντως να κάνουμε και κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά της παράνομης και θα της εργασίας, ε, να έχουμε και ε, κοινούς για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα μαζί ε, σε συνεργασία και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και επίσης να προσπαθήσουμε και με τις χώρες μέλη να έχουμε και κάποιες συστάσεις για να διευκολύνουμε και να λάβουμε υπόψη μα και ότι έχουμε και μικρέ οικογενειακέ γεωργικές εκμεταλλεύσει που και αυτέ πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνε. Αναφερθήκατε επίση και στην εποχική ε, εργασία. Υπάρχουν κάποιε περίοδοι στι οποίε υπάρχει ε, άφθονη δραστηριότητα και ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας και για τον τομέα της γεωργίας ε, διαπιστώσαμε ότι στις χώρες αυτές ε, υπάρχει ε, ευελιξία και υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν κάποιες εποχιακές συμβάσεις και συστήματα εποχιακής εργασίας. Υπάρχουν λιγότερες παραβιάσεις. Για παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχουν ακόμα 38 ώρες την εβδομάδα. Ένας γεωργός εργάζεται 11 ώρες την ημέρα, 50 ώρες την εβδομάδα και να πληρώνει τέτοια ημερομίσθια είναι πολύ δύσκολο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις περιόδους που έχουμε με περισσότερη εργασία, να υπάρχει δυνατότητα συμβάσεων περιορισμένου χρόνου και αυτό βοηθά και τους γεωργούς φυσικά και τις οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις. Και θα απαντήσω και σε μία τελευταία ερώτηση. Ε, νομίζω ο κύριος Καπούτο έθεσε αυτή την ερώτηση. Είπε ότι χρειαζόμαστε παρέμβαση από το δημόσιο τομέα και να υπάρξουν περισσότερα πράγματα από πλευρά κυβερνήσεων. Νομίζω ότι όντω οι χώρε είναι αυτέ οι οποίε μπορούν να παρέμβουν και να δώσουν και κάποιες λύσεις, αλλά όπως είπα, πιστεύω με επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε και τη δυνατότητα στου κοινωνικού εταίρους να συμμετέχουν και να τους ζητήσουμε να βρουν και λύσεις οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Και αν δεν κάνουν τίποτα κοινωνικοί εταίροι, τότε σε δεύτερο στάδιο το Κοινοβούλιο και ε, η κυβέρνηση είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να παρέμβουν. Επίσης αναφερθήκατε και στην ΚΑΠ, ε, αν μπορούμε να έχουμε κάποιους όρους ε, στην ΚΑΠ, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό, διότι Το συζητήσαμε και με τους συναδέλφους της ΖΕΟΠΑ, αλλά εφόσον οι χώρες δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή διάκριση μιας παραβίασης η οποία είναι απλώς μια τυπική διαδικασία και της πραγματικής παράνομης εργασίας, Πιστεύω ότι ένας γεωργός ε, σε μια χώρα, μια μικρή οικογένεια που χρειάζεται κάποιον απλώς για κάποιες εποχιακές δουλειάς, ε, δεν ε, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό ως ε, πραγματική παράνομη εργασία και αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία των ε, παραβιάσεων, των επιθεωρήσεων εργασίας, βλέπουμε ότι δεν γίνεται διάκριση. Και εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ λοιπόν μιας απλής τυπικής παρέβασης και της πραγματικά της εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να αναφερόμαστε σε όρους για την ΚΑΠ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση που σα ανέφερα. Ε, ε, πιστεύω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν έχω ξεχάσει κάτι, ε, θα, παρακαλώ να μου το πείτε, θα μπορέσω να λάβω το λόγο. Να σας ζητήσω όμως το εξή, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή σας. Αναφέρθηκα στην ε, οδηγία για την ε, ασφάλεια στην εργασία, για την κοινωνική ασφάλιση. το γεγονός ότι ο εργοδότης σε κάθε χώρα όταν έχουμε εποχιακούς εργαζομένους σε κάθε χώρα ε, και κάθε χώρα θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας στις χώρες καταγωγής του εποχικά εργαζόμενου, ε, δυσχεραίνουμε πάρα πολύ τη δουλειά των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Σκεφτείτε λοιπόν πώς μπορούμε να τα πλουστεύσουμε, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Είναι ένα θέμα που αποσχολεί τους εργοδότες, το έχουμε συζητήσει και με τα συνδικάτα, συμφωνούν μεταξύ μας. Ε, η Επιτροπή σας λοιπόν, η οποία είναι αρμόδια για να βοηθήσει τη Γεωργία, θα πρέπει να προσπαθήσει να οργανώσει και τα πράγματα ε, με καλύτερο τρόπο, σεβόμενοι και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, σεβόμαστε τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, θα πρέπει να υπάρχουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ε, ε Ασθένειε, να λαμβάνονται υπόψη κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και το να πρέπει να δηλώνονται εκεί πραγματικά αποτελεί πρόβλημα. Σα ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε άλλε ερωτήσει αν ξέχασα κάποια. Σα ευχαριστούμε. Ε, κύριε Πότεχαν, γιατί πραγματικά απαντήσατε διεξοδικά στις ερωτήσεις και μάλιστα χρειάστηκε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο 20 λεπτό σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Μπότερμαν για την συμμετοχή, την παρουσίαση της έκθεσης, τη συμμετοχή στη συζήτηση. Νομίζω ότι διευκρινίσαμε πολλά. Και μάλιστα τη συζήτηση παρακολούθησαν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Μπότερμαν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο Τη ημέρησας διάταξη. Αν υπάρχουν άλλε ερωτήσει μπορείτε να στείλετε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της απορίας σας στον κύριο Μπότερμαν που είναι και πολύ γλώσσος. Οπότε θα σας απαντήσει. Και ευχαριστούμε θερμά και για το υλικό που μας αφέρατε. Πέραμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 11. Όπως θα θυμάστε, Αντί για τη συζήτηση για την κατάσταση της μελισσοκομείας, θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα την παρουσίαση της μελέτης του ΣΤΟΑ με θέμα τη γεωργία ακριβίας και το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη. Το Τμήμα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών ε, εκπονεί διεπιστημονική έρευνα και παρέχει στρατηγικές ε, σύμβουλες στο θέμα επιστήμης και τεχνολογίας, ε, των τεχνολογικών και επιστημονικών επιλογών ε, και κάνει αξιολόγηση και ε, επιστημονικές προβλέψεις. Επίσης, εμβριθείς μελέτες, καθώς και οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για τα θέματα αυτά. Ε, υπό την ίδια της ΤΟΑ, το παρελα... συμμετέχω στο 25 ευρωβουλευτές. Όπως ξέρετε, η κυρία Πετήρο, ο κύριος Νέκοφ και η κυρία Μαγκεντάρ είναι οι δικοί μας εκπρόσωποι, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Γεωργίας στο πάνελ του ΣΤΟΑ. Και μάλιστα θυμάστε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για τη συμμετοχή στην Επιτροπή αυτή. Και μάλιστα έγινε προσπάθεια για αύξηση του αριθμού των ε, αντιπροσώπων κάθε επιτροπής στη ΣΤΟΑ, γιατί πολλοί, πολλές επιτροπές ενδιαφέρονται τα μέλη να παρακολουθούν τις συζητήσεις του ΣΤΟΑ. Η τελευταία ε, μελέτη με θέμα Γεωργία Κρυβίας και το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρώπη διεξήχθη υπό την αιγίδα της κυρίας Μέρετ Μαγκίνες που εποπτεύει αυτά τα ζητήματα ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για την ΣΤΟΑ. Επίσης είναι πολύ δραστήριο μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, μάλιστα, τα γραφεία της κυρίας Μάκενταρ, του κύριο Χαίταμα και του κύριου Ρούμπιχ επίσης ε, παρακολούθησαν ε, και συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης που υπάρχει και ε, ως έγγραφο και ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμη στα μέλη της Επιτροπής. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την Γεωργία Ακριβίας, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο αρμόδιος εμπειρογνώμονας που θα μας παρουσιάσει και τη μελέτη. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και δαπανηρό είναι αυτό το θέμα της ε, γεωργικής παραγωγής και σίγουρα η παραγωγικότητα επηρεάζεται και από την αποτελεσματικότητα των γεωργικών πρακτικών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντεμπερτ Μάκερ για να μας κάνει την παρουσίαση της μελέτης αυτής και του θέματος της γεωργίας ακριβίας. Σας καλωσορίζω και πάλι θερμά και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που μας δίνουν την ευκαιρία να ε, λίγο φως ε, στα θέματα της γεωργίας ακριβίας και το πώς μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη, η γεωργία ακριβίας. Πρόκειται για μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν πολλές αρχές και τη συνοψίσαμε στη συγκεκριμένη έκθεση. Όταν εξετάζουμε τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι 80-85 σχεδόν τα 100 των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερες των 20 εκταρίων. Μόλις 7% είναι μεγαλύτερες από, τα 50, από 50 εκτάρια. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει διαφορά μεγάλη στο μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και η κατανομή τους επίσης είναι άνηση μεταξύ των κρατών μελών. Ένα επιπλέον πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Ένα άλλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της γεωργικής κοινότητας. Μόνο ένας μικρός αριθμός των γεωργών ε, θα συνεχίσουν ε, τις γεωργικές δραστηριότητες μετά από 15 χρόνια. Μάλλον μόνο το 20% των γεωργών αυτή τη στιγμή είναι κάτω των 35 ετών. Οπότε σε 20 χρόνια αυτοί θα είναι οι μόνοι που θα συνεχίσουν ή θα αποτελούν το βασικό τμήμα της γεωργικής κοινότητας. Μόνο το 20% του σημερινού γεωργικού δυναμικού. Οπότε διαρωτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θέλουμε μια παραγωγική γεωργία που θα δίνει ευκαιρίε και στη γεωργική κοινότητα, στους γεωργού και στου νέου γεωργού. Θέλουμε να προσελκύσουμε του νέου γεωργούς, να ασχοληθούν με τη γεωργία για να αποφύγουμε την περίμωση της υπαίθρου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Θα πρέπει να μείνει ο κόσμος στα χωράφια, στην ύπεθρο, στα χωριά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό σήμερα, η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Επίσης, ε, να δούμε τι προβλήματα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη Γεωργία. Μιλούμε για την ε, έξυπνη γεωργική διαχείριση, για την ε, γεωργία της ακριβίας, για την ψηφιοποίηση της κοινωνίας και της γεωργίας, που ίσως μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις μείζονες προκλήσεις του μέλλοντος, που είναι η ασφάλεια των τροφίμων, για τα υγιεινά τρόφιμα, η, περιβαλλοντική ευθύνη και φυσικά και η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η ψηφιοποίηση της κοινωνίας είναι μια πραγματικότητα, ήδη συμβαίνει. Έχουμε τα έξυπνα κινητά, όλοι νομίζω εδώ στην αίθουσα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επίγνωση του πόσο προηγμένη είναι η ψηφιοποίηση αφορά τη βιομηχανία, την καθημερινότητα, το διαδίκτυο των πραγμάτων και ούτω καθεξής η γεωργία ακριβίας μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της ψηφιοποίησης μαζί με κάποια καλή γνώση ώστε να καταλήξουμε στην έξυπνη γεωργία, έξυπνη γεωργική διαχείριση, ώστε να βελτιστοποιήσουμε την ε, γεωργική παραγωγή με συνδυασμό ε, του γονιδιακού χαρακτήρα των καλλιεργιών, της, του περιβάλλοντος, και φυσικά του περιβάλλοντος και του εδάφους σε συνδυασμό ακόμη το καλύτερο, του κλίματος σε όλες τις χώρες και φυσικά και της τεχνολογίας που μπορεί να μας βοηθήσει για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες και όλα αυτά φυσικά με μια χρηστή διαχείριση. Η βελτίωση αυτού του συνδυασμού η βελτιστοποίηση αυτού του συνδυασμού είναι μια μεγάλη πρόκληση. Επίση να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της έξυπνη ε, καλλιέργεια, της έξυπνη γεωρικής ε, διαχείριση. και ποιε είναι οι προκλήσει, Θα πρέπει να γίνονται καταρχήν ε, ακριβείς παρατηρήσει, σωστέ παρατηρήσει. Γιατί όταν πηγαίνουμε στο χωράφι βλέπουμε που υπάρχουν ζυζάνια. Γνωρίζουμε όμω πόσα ζυζάνια, υπάρχουν, μπορούμε να τα καταμετρήσουμε, μπορούμε να δούμε τις ασθένειες, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ε, οι καλλιέργειες ε, λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Και δεν έχουμε μόνο τις ε, παρατηρήσεις, θα, χρειαζόμαστε και σωστή τεκμηρίωση, χάρτες που, του εδάφους και θα πρέπει τέτοια χαρτογράφηση να υπάρχει και να ενημερώνει και για προηγούμενες καλλιέργειες ή τους τρόπους κατεργασίας του εδάφους ε, ή των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν. Όλα αυτά προϋποθέτουν και μια σωστή ανάλυση. Μια σωστή ανάλυση θα μας επιτρέψει να λάβουμε σωστές λύσεις και να ε, επιλέξουμε και το σωστό γονότυπο, γιατί υπάρχουν ε, ποικιλίε σπόρων σιτηρών ή αραβοσίτου που είναι κατάλληλες και συγκεκριμένα εδάφη ή χαρακτηριστικά εδαφικέ διαρθρώσει ε, και προσαρμόζονται σε συγκεκριμένο κλίμα και αποδοκιμούν καλύτερα σε συγκεκριμένε συνθήκε. Οπότε θα πρέπει να στηριχθούμε σε πληροφορίε που δίνουν ε, στου γεωργού οι εταιρείε που πουλούν του σπόρου. Επίση έχουμε πειράματα που ε, βλέπουμε ποια είναι η αξία του κάθε γονότυπου. Όταν έχουμε το γονότυπο, το γονιδιότυπο, γονιδιότυπο που θα πρέπει να το προσδιορίσουμε, θα πρέπει να περάσουμε στη σπορά. Και επίση το θέμα τη εφαρμογή λιπασμάτων είναι σημαντικό. Τι δόση θα εφαρμόσουμε ανάλογα με τον αριθμό των φυτών ανά εκτάριο. Επίσης θα πρέπει να βρούμε τη σωστή δόση του λιπάσματος και να χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα χημικά. Και η χημική σύνθεση του λιπάσματος εξαρτάται από την προηγούμενη ανάλυση που θα έχουμε κάνει για το έδαφος και τα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά του. Και περνάμε στις δράσεις. Θα πρέπει να βάλουμε τη σωστή δόση στο σωστό σημείο για το κατάλληλο φυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και επίσης να φροντίσουμε να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο. Αν ε, γίνει πρόορη σπορά, ε, μπορεί να μην προλάβουμε ε, πολύ καθυστερημένα να χάσουμε την μέγιστη, τη βέλτιστη απόδοση. Επίσης, οι σωστές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες, σωστή πρόβλεψη του καιρού. Και επίσης να έχουμε ε, εύρυθμα λειτουργούσε και καλά προσαρμοσμένε στι ανάγκε μα μηχανέ, γεωργικά μηχανήματα, για να μπορέσουμε πραγματικά να δίνουμε τη σωστή βάση την κατάλληλη στιγμή στο φυτό που χρειαζόμαστε, που θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν διαθεσιμότητα των στοιχείων, τη τεχνολογία και των μηχανημάτων και τη γνώση. Εδώ έχουμε ένα μικρό χωράφι στο οποίο κάναμε κάποια πειράματα αρχικά τα κόκκινα τμήματα είναι εκεί που έχει χάσει χρήματα ο Γιώργος. και ε, αυτά κοστίζουν τα κόκκινα τμήματα και τα πιο σκούρα τμήματα είναι εκεί που μπορεί να έχει κάποιο κέρδος ο Γιώργος. Αν όμως χρησιμοποιεί χημικά και λιπάσματα ομοιόμορφα σε όλο το χωράφι δεν έχει νόημα. Οπότε μπορεί να βελτιωθεί από αυτή την άποψη η διαχείριση. Και εκεί ερχόμαστε στην ε, γεωργία ακριβία. στη διαχείριση των ε, κλιμάκων μεγέθους και των προσεγγίσεων. έχουμε μια εφαρμογή σε επίπεδο αγρο, αγρού και παίρνουμε μερικά δείγματα εδάφους ανά εκτάριο ή ανά πέντε εκτάριο και θεωρούμε ότι έχουμε τις σωστές πληροφορίες για το σύνολο του αγρού. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι σωστό γιατί υπάρχουν διαφορές στην υφή του εδάφους και στις ηθίκες του εδάφους και στην κατάσταση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Στην γεωργία ακριβίας λοιπόν υποδιαιρούμε τον αγρό ε, σε επιμέρους αγροτεμάχια, σε επιμέρους ε, περιοχές, ώστε εκεί που χρειάζεται λιγότερο λίπος με λιγότερο φυτοφάρμακο να έχουμε λιγότερη εφαρμογή και σε άλλες περιοχές μπορούμε να περιορίσουμε το, τη δόση των λιπασμάτων γιατί ούτως ή άλλως δεν βοηθά να έχουμε αυξημένη παραγωγή εκεί. Το ίδιο ισχύει και για τα ζυζανιοκτώνα ή για τον έλεγχο των εχθρών των φυτών και των επιβλεβών οργανισμών. Και σίγουρα στο μέλλον δεν θα έχουμε μόνο ειδική διαχείριση ανά τμήμα, αλλά και ε, θα μιλούμε για διαχείριση μεμονωμένων φυτών και δέντρων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γιατί και η απόδοση και η ποιότητα της συγκομιδής ε, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Οπότε μπορούμε να μιλούμε για την τεχνολογία και έχω κάποιες διαφάνειες για το θέμα αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ποιος είναι και ο αντίκτυπος της γεωργίας ακριβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών θα συμβάλλει, πιστεύω, σημαντικά στην ασφάλεια και την προστασία των τροφίμων. Ίσως εδώ η τεχνολογία της έξυπνης καλλιέργειας και της γεωργίας ακριβίας μας επιτρέπει με λιγότερα μέσα, με λιγότερες ροές να έχουμε ε, μεγαλύτερη παραγωγή. Δηλαδή, μεγαλύτερη παραγωγή με μικρότερες χημικές ή άλλες γεωργικές ροές ή να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων σε λιγότερη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας το έπακρο τα πιο γόνιμα τμήματα, τα πιο γόνιμα εδάφη. Αν το καταφέρουμε λοιπόν, θα προωθήσουμε ταυτόχρονα και την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των φυτών, γιατί θα χρησιμοποιούνται λιγότερα φυτοφάρμακο. Επίσης υπάρχουν, ε, είναι και πιο αηφόρος ο τρόπος αυτής της γεωργίας, της γεωργίας ακρίβειας και σε μερικές περιπτώσεις έχουμε και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Και σημαντικά ωφέλη και στην παραγωγικότητα και κέρδη εκεί στην παραγωγικότητα. Επίσης, είναι και θέμα κοινωνικών αλλαγών. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών θα πρέπει να αυξηθεί και ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές, ώστε ε, να έχει κάποιο γόητρο η γεωργία και να μην είναι μόνο χειρονακτική εργασία, αλλά να είναι και διανοητική και τεχνολογική πρόκληση. Επίσης, πώς επηρεάζονται οι εργασιακές πρακτικές και οι ε, βιωτικές συνθήκες της γεωργικής εκμεταλλεύσης ε, ή να επιτρέψει οι Γιώργος να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και κοινωνικέ δραστηριότητε ή να δημιουργηθούν νέα επιχειρησιακά γεωργικά μοντέλα για να αυξηθεί καλύτερα η κατάρτιση και στη διαχείριση των δεδομένων, άλλο σημαντικό τμήμα της βελτίωσης αυτής της, της γεωρικής πρακτικής. Θέλουμε λοιπόν φυσικά και νέες δεξιότητες, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, αλλά και διαχείρισης, διαχειριστικές. Όλες αυτές απαιτούνται για, το, για την έξυπνη, για τη γεωργία ακριβίας. Είναι πρόκληση λοιπόν αυτό για τους νέους ε, αγρότες, αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία γιατί αυτή τη στιγμή το αγροτικό εισόδημα κατά μέσον όρο είναι κατώτερο το υπολείπο εισοδήματος της κοινωνίας. Άρα θα υπάρχει και ένα κοινωνικό ε, στάτους, ένα γόητο να εργάζεται κανείς στη Γεωργία. Η γεωργία ακριβίας όμως θα πρέπει να είναι και προσιτή και εφικτή ανεξαρτήτως είδους γεωργικής εκμετάλλευσης ή μεγέθους. Μπορεί να υπάρχει η μεγάλη υπαρχει καλλιέργεια σιτηρών, ας πούμε, ή μικρή με καλλιέργεια οπωροκυπευτικών και να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, όχι όμως στο παραδοσιακό κλάδο της γεωργίας, αλλά σε τομείς δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στη γεωργία. Όλα αυτά είναι πρόκληση και για εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαράσουν τις πολιτικές. Οι ευκαιρίες της γεωργίας ακριβίας εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την απόψή μου. Λοιπόν, για να προσπαθήσω να συνοψίσω. Τι είναι η γεωργία ακριβίας. Συγκέντρωση δεδομένων, παρακολούθηση, ανάλυση, ε, καθοδήγηση της παραγωγής και διαχείρισή της. Παράγουμε περισσότερα με λιγότερα και εκμεταλλευόμαστε ε, την ποικιλία των εδαφών και του κλίματος. Βεβαίως όλα αυτά συνδέονται με τα δεδομένα, εξαρτώνται από την τεχνολογία, αλλά και από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Ήπεθρο και στις αγροτικές κοινωνίες, κοινότητες. Βασίζεται στην πληροφορία, βασίζεται στη γνώση για τη λήψη των αποφάσεων. Με τα λόγου γνώσεως λαμβάνεται η δράση ε, για όλα τα είδη γεωργίας και απασχόλησης. Σήμερα οι γεωργοί έχουν την πίεση να αποδείξουν και την υποχρέωση ότι χρησιμοποιούν ορθές γεωργικές πρακτικές. Στις τεχνολογίες ε, γεωργίας ακριβίας αυτά παράγονται αυτόματα ως στοιχεία και αυτό ε, διευκολύνει ε, τη δυνατότητα που έχουν οι αγρότες να ε, πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με όλα αυτά που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν η γεωργία ακριβίας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Παράδειγμα, πρόληψη της διάβρωσης, πρόληψη των πλημμυρών, ε, βέλτιστη χρήση ε, των ε, λιπασμάτων και ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα. Τα υπόγεια ύδατα προστατεύονται από τη διαρροή αζότου, από τα νητρικά ε, μειώνονται τα χημικά για την προστασία των φυτών, καλύτερη διαχείριση των ζυζανίων, το ίδιο ισχύουν και εδώ. Και άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμα και με τη χρήση λιγότερων χημικών μπορούμε να μειώσουμε τις ζημιές από επιβλαβείς οργανισμούς ή από μύκητες που προσβάλλουν τα φυτά. Επίσης, ε, μπορούμε να έχουμε άμυψη σπορά ή μικτές καλλιέργειες για να ε, τονώσουμε τη βιοπικιλότητα και να βελτιώνουμε τα εδάφη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ε, καλή δομή του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, για τη διατήρηση της καλής ποιότητας των εδαφών μας. Η γεωργία ακριβίας ε, ενδεχομένω να έχει και επιπτώσεις για την κοινή γεωργική πολιτική. Η ενίσχυση του εισοδήματος, η ενίσχυση ε, της εφαρμογής και της ανάπτυξης ε, της γεωργίας ακριβίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί η επίπτωση στον περιβάλλον, να έχουμε Υψηλή τεχνολογία καλλιέργειε που να σέβονται το περιβάλλον και να είναι φιλικές και προ την απασχόληση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την μετατροπή των καλλιεργειών σε καλλιέργειε ε, ακριβία με τεχνικές εφικτέ. Δεν χρειάζονται πάντα πολύ μεγάλα γεωργικά μηχανήματα και περίπλοκα. Ε, μπορεί να γίνει αυτό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ε, θα πρέπει να ασκείται αυτή η γεωργία Ακριβία ε, από εκπαιδευμένου αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέε δεξιότητε και επιχειρηματικές και διαχείρισης δίκης επιχειρήσεων και ανεξαρτήτως του μεγέθους της εκμετάλλευσης. Υπάρχουν και άλλοι τομεί πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η γεωργία Ακριβία μπορεί να έχει επιπτώσεις ή να επιπτώσει η περιβαλλοντική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, γιατί Έχουμε ε, εναλλακτική απασχόληση, πολιτική ανταγωνισμού, καινοτομία και επιστήμη, ψηφιακή πολιτική στην εποχή της ψηφιοποίησης και τι γίνεται με την ιδιοκτησία των δεδομένων. Αυτό είναι ακόμα υποσυζήτηση. Και βεβαίως εδώ χρειάζεται εκπαίδευση και κατάρτιση ε, στην Ήπεθρο και να αλλάξουν οτροπία και οι εκπαιδευτές. Ε, των αγροτών. Επίσης στην ε, βιομηχανική πολιτική, ακόμα και οι κατασκευαστές δηλαδή γεωργικών μηχανημάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ε, θα σταματήσω εδώ για ερωτήσει. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σα δώσω και κάποια ακόμα παραδείγματα, αλλά νομίζω κατά τη συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε πραγματικά την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί δεν έχουμε πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη. Μάλιστα, ο καλεσμένος μας είναι καθηγητής ε, Πανεπιστημίου και χαίρομαι που βρήκε χρόνο για συζήτηση μαζί μας. Στην οποία θα περάσουμε τώρα. Κύριε Νόεχλου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο. Θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα επόμενα έτη αλλά και δεκαετίες ολόκληρες. Είπατε ότι για τη μικρή και μεγάλη γεωργία υπάρχει δυνατότητα γεωργία ακριβίας. Εγώ θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Πώς είναι δυνατόν οι μικροί αγρότες να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Υπάρχουν αγρότες που δεν είναι αγρότες σε κατά κύριο επάγγελμα. Πώς μπορεί κανείς να ακολουθήσει εξελίξεις και μόνο από το τεχνικό εξοπλισμό και πώς να ανταγωνιστεί με τη μεγάλη γεωργία. Αυτό ευνοεί τη μεγάλη γεωργία. Επίσης είπατε ε, να παράγουμε περισσότερο με λιγότερα εφόδια. Εδώ ο λογαριασμός βγαίνει μόνο κατά το ίμιση γιατί τα προϊόντα που χρειαζόμαστε ε, και τα μηχανήματα και τα λοιπά είναι και αυτά σε μια διαδικασία παραγωγής και θα πρέπει να παραχθούν. Δεν μπορούμε να υποδιόμαστε ότι τελικά αυτό είναι βελτίωση με λιγότερη ενέργεια ή με λιγότερα εφόδια για να έχουμε περισσότερη παραγωγή. Νομίζω δεν έχετε λάβει όλες τις παραμέτρους υπόψη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος παραγωγής των ε, γεωργικών μηχανημάτων. Και κάτι ε, που είναι για μένα πιο σημαντικό και πιο δύσκολο είναι κάτι που το πνίξατε λίγο, γιατί όσο περισσότερη τεχνολογία, τόσο περισσότεροι ε, εργαζόμενοι. Τι γίνεται με την γραφειοκρατία, παρουσιάσατε ε, έναν αγρότη που θα αλλάξει επάγγελμα στο μέλλον. Πρέπει να είναι και λίγο χημικός, πρέπει να είναι και λίγο ε, ε κομπιουτεράς. Είναι δυνατόν οι περισσότεροι αγρότες να υποφεληθούν. Αυτό θα ευνοήσει μόνο ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα των σημερινών γιώργων. Μα δεν θα έχει άλλη Ο κύριος Βαλκάρσελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και πολλοί από εσά, αν όχι όλοι, γνωρίζετε ότι είμαι μέλο ε, τη της Επιτροπή αυτή ω αναπληρωτή, αλλά ω αντιπρόεδρο είμαι αρμόδιο εξ ονόματο του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούν την Επιστημονική Επιτροπή ΣΤΟΑ. Και η Επιτροπή αυτή είναι αυτή η οποία προσφέρει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητες ποιοτικέ πληροφορίες για τον αντίκτυπο των ε, προόδων ε, της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών ε, και τι μπορούν να προσφέρουν στα θέματα που μας αποσχολούν. Και φυσικά ε, διαθέτουν σε όλους τους ευρωβουλευτές τα συμπεράσματα και τις συστάσεις ε, των επιστημονικών μελετών ε, ιδιαίτερα αυτών που είναι γνωσμένου κύρος, ώστε να μπορέσουν να τα λάβουν υπόψη τους όταν αξιολογούν και καθορίζουν στρατηγικές πολιτικές ε, βράχη, πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεισφοράς της ε, στις ε, κοινοβουλευτικές εργασίες, η ΣΤΟΑ παρουσιάζει πολύ σημαντικές μελέτες όπως αυτή που μόλις ακούσαμε από τον καθηγητή για την γεωργία ακριβίας και το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη που θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω, αν μου επιτρέπετε, ότι η Μούρθια, η περιοχή καταγωγής μου, ε, ζει σε μεγάλο βαθμό από την πλήρη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων που ε, είναι και ε, σπάνιοι και σε ορισμένες περιπτώσεις πρακτικά ανύπαρκτοι. Η γεωργία Κρυβίας λοιπόν είναι η μεγάλη σύμμαχος αυτής της περιοχής ε, η οποία έμαθε να δίνει μάχες ε, κατά ενός πάρα πολύ ξηρού ε, κλίματος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Για παράδειγμα αναπτύσσοντας την βέλτιστη προετοιμασία του εδάφους εγκαθιστώντας αυτοματοποιημένα συστήματα ε, ποτίσματος και άρδευσης και φυσικά ε, και πάρα πολλές άλλες τεχνικές οι οποίες υποβοηθούν τις διαδικασίες. Μέσω λοιπόν των πολύ σημαντικών επενδύσεων σε καινοτομία και έρευνα η ε, κυβέρνηση της αυτόνομης περιοχής τα, τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε μεγάλη όθηση στην γεωργία ακριβίας. Όλα αυτά επέτρεψαν ε, στη Μούρθια να γίνει μία από τις ε, πρωτοπόρες ε, περιοχές στην εκμετάλλευση αυτών των καινοτομιών και μπόρεσε φυσικά να εξοικονομήσει και να χρησιμοποιήσει με κατάλληλο τρόπο τους υδάτινους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Και φυσικά αυτό βοήθησε ιδιαίτερα. Ελπίζω λοιπόν η μελέτη τη ΤΟΑ να βοηθήσει όλου να εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητε που προσφέρουν αυτέ οι τεχνολογίε, οι οποίε προσαρμοσμένε στι κατάλληλε ε, ανάγκε τη κάθε περιοχή θα μπορέσουν να βοηθήσουν να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των περιοχών τη υπαίθρου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε Πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε. Γιατί έτσι διευρύνεται και τον ορίζοντα των γνώσεών μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Ντενανό. Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι επανειλημμένα η Επιτροπή μας έχει προβληματιστεί για ε, αυτό το θέμα της ε, γεωργίας ακριβίας. Είχαμε και την έκθεση του συναδέλφου Χάιτεμα ε, που πραγματεύεται αυτά τα θέματα. Κύριε καθηγητά, είπατε στόχος είναι να παραμένει ο κόσμος στην Ήπεθρο και είναι πάρα πολύ αξιέπαινος αυτός ο στόχος. Δεν θα πρέπει ε, να το λησμονούμε αυτό, βεβαίως ε, να αποφεύγουμε σπατάλες και να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Ε, θα πρέπει να έχουμε συλλογή πληροφοριών για τη σύσταση των εδαφών, για τη γεωργική κατάσταση, του, γεωγραφική κατάσταση, το κλίμα, τι μετρολογικές συνθήκες και με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους για να προχωρούμε και να δούμε ποιο θα είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό και οι σπόροι που θα χρησιμοποιούνται εκεί στα διάφορα εδάφη. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα πολλές φορές και το είπε και στην Άρφος Νόχελ. Οι μικροί αγρότες μπορούν να απαντήσουν σε όλα αυτά τα πολύ επιστημονικά ερωτήματα. Αυτά είναι ανέφικτα πράγματα για τους παλιούς. Τώρα από την άλλη νέοι αγρότες, η νέα γενιά είναι πιο πολύ εξοικειωμένοι και με την πληροφορική και με την γεωστρατηγική. Ε, θα πρέπει ε, πραγματικά να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και να προβληματιστούμε γιατί μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτή την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να είναι ηγετική σε αυτή την προσπάθεια και το χαιρετίζω. 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε γράψει ε, στο πρόγραμμα Horizon 2020 ακριβώς για αυτό το θέμα, για τη γεωργία ακριβίας. Και ε, πρέπει να έχουμε απολύτως επίγνωση ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις καταστάσεις και με βάση τις προτάσεις που κάνετε, που είναι ενδιαφέρουσες, να προχωρήσουμε στην πρότασή μας για τη νέα ΚΑΠ, να εισακάγουμε αυτή την ιδέα ε, του ε, αγρότη επιστήμονα ε, για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση θα μας βοηθήσει πολύ στις συζητήσεις μας με τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών. Γιατί αυτή την απόφαση λάβαμε με τους συντονιστές. Να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών. Πρόκειται για μια διεύθυνση που συντονίζει τις μελέτες ε, για θέματα καινοτομίας ε, και άλλα. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γεωργία ακριβίας ε, αναμφισβήτητα αποτελεί στρατηγικό μέσο για το μέλος, ε, μέλλον συγγνώμη, της γεωργικής εκμετάλλευσης ε, με βάση φυσικά και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ρομποτική, τα ντρόουν, οι δορυφόροι είναι εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν να μειώσουμε αισθητά τη χρήση φυτοφαρμάκων, υδάτινων πόρων, ορυκτών καυσίμων και επίσης ε, θα συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση της απασχόλησης των νέων, δεδομένου ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες απαιτούν και ε, ψηφιακές γνώσεις, τις οποίες μόνο οι νέοι μπορούν να εξασφαλίσουν. Αυτή είναι η ε, καλή πλευρά της ε, Γεωργίας Ακριβίας και από αυτή την πλευρά θα έλεγα ότι η μελέτη της ΣΤΟΑ δείχνει με σαφή τρόπο όλα αυτά τα ε, στοιχεία και όλες αυτές τις δυνατότητες. Το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε ε, στους εαυτούς μας περισσότερο και όχι σε εσά, ε, εμείς που είμαστε πολιτικοί θύνοντες, είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τις νέους τρόπους γεωργίας χωρίς να ζημιώσουμε και τις περιοχές της υπαίθρου και τρόποντινά και τις μικρές εκμεταλλεύσεις ε, όπως αναφέρθηκε, διότι ο πραγματικός κίνδυνος που ελοχεύει είναι να έχουμε περαιτέρω περιφερειοποίηση των ε, μικρών, πάρα πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων που τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο ε, της έναρξης αν θέλετε του startup, δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ε, τους κολοσσούς του γεωργικού κλάδου. Και από αυτή την άποψη, όπως έλεγε και ο προλαλής σας συνάδελφος, η νέα ΚΑΠ θα πρέπει ε, να έχει όλο ένα και πιο συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξει και ε, την κατάρτιση των νέων γεωργών και να βοηθήσει και την ε, ψηφιακή γνώση στις περιοχές της υπαίθρου. Πολύ συχνά ε, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα, δεν επενδύουν στις περιοχές της υπαίθρου ακριβώς γιατί είναι λίγα λίγοι μάλλον οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση τη μελέτη. Σε μερικά σημεία έχω απογοητευτεί λίγο για το αποτέλεσμα, για το πώς αξιολογείται αυτό όταν διαβάζω την έκθεση βλέπω ότι υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Ας πούμε αριθμός και μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην πρωτογενή παραγωγή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν βλέπω πώς περιορίζεται η ανεργία των νέων. Μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών. Αλλά αν κοιτάξω τι γίνεται στην πράξη, και ότι θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους στην Ήπεθρο, βλέπουμε νέους που θέλουν να επιστρέψουν στην Ήπεθρο, να αρχίσουν μια γεωργική εκμετάλλευση με γεωργία ακριβίας. Αυτοί το κάνουν ε, μαθαίνοντας τις μεθόδους καλλιέργειας, τις βιολογικές καλλιέργειες και με άλλους τρόπους διάθεσης των προϊόντων στην ε, αγορά. Πώς θέλετε να κρατήσετε τους νέους με περισσότερη τεχνολογία στην Ήπεθρο, τολμώ να το αμφισβητήσω. Έχουμε τεχνολογία ήδη στις εκμεταλλεύσεις, δεν είναι αυτό που λείπει. Αυτό που λείπει είναι το εισόδημα, αναφερθήκατε σε αυτό, είναι κάτω από το μεσόωρο και αυτό μπορεί να λυθεί με παραγωγή μεγαλύτερης ακριβίας. Τολμώ και αυτό να το αμφισβητήσω, αν δεν είναι εντάξει αγορές. Το πρόβλημα δεν είναι πώς παράγουμε. Μια χαρά παράγουμε, αλλά όταν χαμηλές οι τιμές διάθεσης, τι να την κάνω την γεωργία ακριβίας. Και το ίδιο ισχύει με το κοινωνικό καθεστώς. Γιατί να έχουν μεγαλύτερο γόητρο οι αγρότες με περισσότερη τεχνολογία. Και αυτό τολμώ να το αμφισβητήσω δεν είναι τόσο κακή η κοινωνική θέση, η αναγνώριση από την κοινωνία ε, των αγροτών, αν παράγουν με τρόπους που να αποδέχεται ο κόσμος. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν τεχνολογία, αλλά αποδοχή στα μάτια του πληθυσμού για αυτά που κάνει η Γεωργία. Ε, λιγότερα ζυζανιοκτώνα, ναι, λιγότερα χημικά και φάρμακα, ναι. Αυτό γίνεται με γεωργία ακριβίας ή με καλύτερες γνώσεις των αγροτών και των αγροτησών για το τι συμβαίνει ε, σε μια καλλιέργεια, τι συμβαίνει στο έδαφος, το υπέδαφος. Ποιος μαθαίνει για τη ζωή του εδάφους, τι γίνεται μέσα στο έδαφος, πώς εξηγιένεται το έδαφος Πουθενά σχεδόν δεν διδάσκεται αυτό. Και εσείς θέλετε να τους βάλετε να μαθαίνουν υπολογιστές και τεχνολογία χωρίς να ξέρουν ε, πώς αλληλεπιδρούν ε, τα φυτά, ποια είναι μια καλή σπορά, πώς δηλαδή πρέπει να διαδέχονται οι καλλιέργειες μία την άλλη. Αυτά δεν τα μαθαίνουν οι αγρότες. και δεν είναι ομοιογενέ το έδαφος ένα αγρόκτημα. Κοιτάξτε, οι παλιοί αγρότες πώς καλλιεργούσαν, είχαν ένα χωράφι και ήξεραν πάρα πολύ καλά ε, ποιο κομμάτι του αγρού προσφέρεται για ποια καλλιέργεια και ποιο λιγότερο και ποιο ε, κομμάτι θα καλλιεργούσαν και θα εκμεταλλεύονταν με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τα ήξεραν πολύ καλά και τον αγρό τους γιατί πατούσαν στο έδαφος. Τώρα κάθονται σε ένα τρακτέρ 2,5 μέτρα από το έδαφος και δεν έχουν επαφή ε, με τη γη και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Ο αγρότης θα πρέπει να ξέρει τη γη του ε, από τη δική του παρατηρήση, από τη δική του γνώση και αν υπάρχουν και κάποια δεδομένα τεχνολογικά να τον υποβοηθήσουν καλώς. Αλλά τώρα απλώς να συλλέγουμε δεδομένα, να τα αξιολογούμε και να κάνουμε αυτό που μας λέει η αξιολόγηση χωρίς να ξέρουν οι αγρότες τι συμβαίνει στο χωράφι τους, δεν πρόκειται καθόλου να προχωρήσουμε. Ούτε στο περιβάλλον, ούτε στο κλίμα, ούτε πουθενά. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούν ε, τα κομπιούτερ. Θα τους λέει το κομπιούτερ τι είδους ε, και τι χαρακτηριστικά έχει το έδαφος θα είναι χρήσιμο αυτή την άποψη. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Εγώ δεν είμαι τόσο επικριτική όσο η προλαλή σα. Δεν τα βλέπω τόσο μαύρα, γιατί στη μελέτη σας πιστεύω αξιολογήσατε και μελετήσατε και τους κινδύνους και τα ε, όρια και τα καταδείξατε. Αρχίσατε από τη δομή διοίκηση των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί το 21% ε, είναι μόλις ε, είναι κάτω από τα 44 και 54% άνω των 55. Αυτά είναι οι ηλικίε των τυχεοργών και δεν ξέρω κατά πόσο η παλιότερη γενιά μπορεί τώρα πια να μάθει, πόσο μάλλον να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για τη γεωργία ακριβίας. Βεβαίως να υπάρχουν τα δεδομένα ασφάλεια του διαδικτύου, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα για μένα, που θα παίξει όλο και περισσότερο ε, ρόλο και η τεχνολογία, ξέρετε, είναι ακριβή. Η τεχνολογία για τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να πω ότι έχουν δίκιο κάποιοι προλαλήσαντες. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, ενώσεις παραγωγών που μοιράζονται τα ίδια μηχανήματα, αλλά τελικά ποιος βγάζει λεφτά, η τεχνολογία, η βιομηχανία, αυτοί που παράγουν ε, ελκυστήρες και δεν έχουμε προστιθέμενη αξία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες, αλλά αν κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, ε, τι διαφορές ε, κρατούν από χώρα σε χώρα και ποια είναι η αποδοχή ε, μεταξύ των γεωργών στη βάση. Δεν είναι δεδομένη. Ούτε το επίπεδο εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ίδιο. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Και τελικά η φύση δεν μπορεί να προγραμματίζεται μέχρι τελευταίας ε, λεπτομέρειας. Κοιτάξτε ε, τι έγινε με τις διάφορες ε, θεομηνίες και τα ακραία φαινόμενα στα κράτη πρόσφατα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να ενταθεί η εκπαίδευση των γεωργών, αλλά να δούμε εμείς ποιες συνέπειες ε, θα έχουμε και ποια συμπεράσματα θα βγάλουμε για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Πώς θα ενισχύσουμε τη μικρή γεωργία. Γιατί η γεωργία σήμερα δεν είναι ενιαία. Πολλές φορές οι καταναλωτές έχουν άλλες επιθυμίες από ε, τους παραγωγούς και οι καταναλωτές καμιά φορά παραπλανώνται και παραπληροφορούνται από τηλεοράσεις, μίντια, διαφημίσεις κλπ. Ε, γεωργία ακριβία, πώ γίνεται με τεχνολογία, με μεγαλύτερου ελκυστήρε, με μεγαλύτερα μηχανήματα. Και αυτό είναι κάτι καλό και για το περιβάλλον. Όλα αυτά πώς θα τα εξηγήσουμε. Και αν δούμε τις ιδεολογικές συζητήσεις που γίνονται στη Γερμανία, δεν θα τα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε ως κάτι θετικό την γεωργία ακριβίας που να εξοικονομεί τους πόρους, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον να ε, ε, το σέβεται. Χαίρομαι που όλοι ενδιαφερόμαστε και ανησυχούμε για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να το λάβουμε εγώ στη συζήτηση του περιπολογισμού για την κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί Εκεί δεν συμφωνούμε ούτε καν στην Επιτροπή μας να στηρίξουμε με τα επαρκή κονδύλια τις ε, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε με τους μικροκαλλιεργητές. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ε, εντατικής καλλιέργειας. Είναι όμως ε, ανάμεκτη κατηγορία αυτή. Μερικές φορές και μικροκαλλιεργητές ε, ασχολούνται με την εντατική γεωργία, γιατί μερικές φορές συναισθηματικά κάνουμε διάκριση μεταξύ μεγάλων καλλιεργητών εντατικής καλλιέργειας και μικρών που είναι εξορισμού εκτατική. Δεν ισχύει αυτό. Επίσης, η έκθεση αυτή αφορά το μέλλον και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτό θα είναι το μέλλον άσχετα από τι πρεσβεύουμε εμείς. Ήδη τέτοιε εξελίξει λαμβάνουν χώρα και μονομένε αγροτικές εκμεταλλεύσει ήδη υιοθετούν αυτές τις τεχνολογίες. Γιατί όμως η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι χαμηλή, γιατί ε, δεν είναι εξίσου ενθουσιώδης υπέρ της γεωργίας ακριβίας όλοι οι γεωργοί. Είπατε ότι απαιτούνται νέες δεξιότητες. Τα κράτη-μέλη έχουν επίγνωση, οι γεωπονικές σχολές, τι ε, ε, τις ανάγκες της του, του προγράμματος, του διδακτικού, προκειμένου να ε, γίνεται καλύτερη κατάρτιση πια και των γεωπόνων και των μελλοντικών γεωργών. Επίσης, μας δείξατε από τις διαφάνειες ότι σε κάποια τμήματα, σε κάποια αγροτεμάχια, ο γεωργό ζημιώνεται και στην κοινή γεωργική πολιτική έχουμε κάποια μέτρα οικολογικοποίηση, πρασινίσματος. Γιατί λοιπόν αυτά τα ε, σημεία του πρασινίσματος να μην αντιμετωπίσουμε σαν τις κόκκινες περιοχές και ίσως στο μέλλον, στη συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τις δεξιότητες που επισημάνατε ότι χρειάζονται στην έκθεσή σας. Το ίδιο ισχύει και για τις μηχανές. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα μηχανήματα, αλλά μηχανήματα που θα είναι διαφορετικά από τα μηχανήματα του παρελθόντος, θα είναι πιο εκλεπτισμένα, πιο περίπλοκα και θα ευθυγραμμίζονται με τις ε, γεωργικές ισορροές. Επίσης, πώς θα αντιδράσει η βιομηχανία παραγωγής φυτοφαρμάκων στις προτάσεις, γιατί θα χρειάζονται πια λιγότερα φυτοφάρμακα στο μέλλον. Θα χρειάζονται λιγότερες ζωικές ισορροές σε επίπεδο φυτοφαρμάκων, αν έχουμε καλύτερη στόχευση. Και κάτι τέτοιο θα επηρεάσει και την, ε, τους παραγωγούς ε, γεωργικών ισρών και δι φυτοφαρμάκων. Και τέλος, κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει η δική μας Επιτροπή με τις πληροφορίες που μας παρέχεται, γιατί όταν η ΣΤΟΑ εκπονεί μια πολύ ουσιαστική μελέτη σαν αυτή, καλό θα ήταν να μην μείνει ξεχασμένη σε ένα σιρτάρι, αλλά να εφαρμοστεί. Τι καθοδήγηση θα μπορούσατε να μας δώσετε, τι κατευθυντήρες γραμμές ώστε να εφαρμόσουμε και εμπράκτος τα πορίσματα της μελέτης σας. Ευχαριστώ κύριος Νέκοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά, είμαι μέλος της ΤΟΑ και με ενδιαφέρει ιδιαίτερως η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την γεωργία ακριβίας. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα φυτοφάρμακα με τα βιοφυτοφάρμακα. Δηλαδή ε, τα ζενιοκτώνα ε, που ή τα παραστοκτώνα που δεν ε, επηρεάζουν αρνητικά το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα ή πώς θα καταπολεμήσουμε επίσης τη διάβρωση του εδάφους. Γιατί οι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την ε, βελτίωση των αποτελεσμάτων αλλά και για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και για την καταπολέμηση της ε, διάβρωσης του εδάφους. Συμφωνείτε μαζί μου? Κύριε καθηγητά, θαυμάζω την απόλυτη πίστη σας στην τεχνολογία και την τεχνική. Ότι πιστεύετε ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του μέλλοντος βασιζόμενοι αποκλειστικά στην τεχνολογία και την τεχνική. Τα προβλήματα των Ευρωπαίων αγροτών δεν είναι ότι δεν παράγουν αρκετά. Το αντίθετο. Υπερπαραγωγή, έχουμε πλεονάσματα. Κοιτάξτε τι γίνεται στα γαλακτοκομικά. Τι θέλει τώρα μεγαλύτερη ακρίβεια για να παράγουμε περισσότερο γάλα. Και πού θα το πάμε. Και δεν πιστεύω και την θέση που λέει και την άποψη ότι τελικά θα χρησιμοποιούνται λιγότερα λιπάσματα και λιγότερα χημικά. Όταν βάλουμε σε ένα ακριβό μηχάνημα τον αγρότη δεν θα περάσει μια φορά πάνω από το χωράφι, αλλά και δυο και τρεις, γιατί θέλει να αποσβέσει και το μηχάνημα. Δηλαδή και θα το ραντίσει τρεις φορές αντί για μία. Η περισσότερη τεχνολογία σημαίνει και περισσότερη χρήση αυτής. Και δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερη η τεχνολογία. Ε, όταν έχεις τη τεχνολογία, το χρησιμοποιείς. Όταν το αυτοκίνητό σου δεν καίει πολύ, δεν το χρησιμοποιείς λιγότερο ή θα κάνεις λελογημένη χρήση, αλλά περισσότερο ακριβώ επειδή δεν καίει. Δεν αναφέρεται κανένα κίνδυνο. Λες και είναι τελείως ακίνδυνη όλη αυτή η τεχνολογία. Και ρωτώ, και ποιος θα τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά. Η απάντηση βρίσκεται λίγο πιο κάτω στη μελέτη σας. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική, λέει, θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσει. Ωραία. Ε, ε, και ποιο θα υποφεληθεί, γιατί ένα ευρώ μπορεί μία φορά μόνο να το δαπανίσει. Ε, και ποιο θα υποφεληθεί οι κατασκευαστέ αυτών των μηχανημάτων και όχι ο Γεωργό. Αυτοί που παράγουν τα μηχανήματα και τα διαθέτουν στην αγορά. Δηλαδή νέε τεχνολογίες, νέε βιομηχανίες και τελικά δεν πάει στην τσέπη του αγρότη αλλά στην τσέπη του βιομηχάνου στη δεκαετία του 60 και του 70 το έχουμε ξαναζήσει που πιστεύαμε ότι όλα θα λυθούν από την τεχνολογία. Δεν τα πιστεύω αυτά. Και εσείς έχετε σαφέστατο αίτημα να έρθει να τα πληρώσει η κοινή γεωργική πολιτική γιατί αυτή είναι η γεωργία του μέλλοντος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ε, είναι αποδοτικό για ε, την ε, πλειονότητα των αγροτών. Και ένα άλλο ερώτημα που δεν απαντήσατε ε, είναι ένα που παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη νέα τεχνολογία. Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα. Είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα και πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες δεν τα συλλέγουν, τα βρίσκουν κάπου αλλού τα δεδομένα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που τα διαχειρίζονται και ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες. Και δεν είναι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι διοκτήτες εκεί. Αυτό είναι πρόβλημα. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα δεδομένα. Στη χημική βιομηχανία που δίνει μια συμβουλή στον αγρότη για πώς θα χρησιμοποιεί τα λοιπάσματα. Όταν μιλάμε για τη διάθεση των δεδομένων, τίθεται και το θέμα της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των δεδομένων. Δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό. Και σε μια σοβαρή συζήτηση ανήκουν και αυτά τα θέματα. Για να το ξεκαθαρίσω, μην νομίζετε ότι εγώ είμαι εχθρός τεχνολογίας. Το αντίθετο να την αξιοποιούμε, να τη χρησιμοποιούμε όπου γίνεται αυτό. Αλλά δεν συμφωνώ καθόλου ότι είναι η λύση όλων των προβλημάτων όπως το παρουσιάσατε. Δεν είναι δυνατόν. Ε, ε, κατά ένα τμήμα ναι, αλλά να μην επενδύσουμε εκεί τα μελλοντικά κονδύλια από την κοινή γενική ε, γεωργική πολιτική, γιατί νομίζω θα είναι αναθασμένη αυτή η απόφαση. Κύριε Ευρωβουλευτά, δεν είναι σωστό ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η γενίκευση της χρήσης της ε, οδηγεί σε μείωση του κόστους και άρα αυξάνει την προσβασιμότητα και μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες οικονομίες ε, που μπορούν να επανεπαιδηθούν στη χρηματοδότηση της επιχείρησης ή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Προσπαθήσαμε να και μια διαφορετική σκοπιά στο πρόβλημα αυτό. Ε, ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα αυτά που είπε ο Μάρτιν Χόισλινγκ πριν από λίγο. Και έχω την εντύπωση ότι συζητούμε αν η τεχνολογία αυτή θα έρθει ή δεν θα έρθει. Μα δεν είναι αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον δεν εξαρτάται από εμά. Φυσικά υπάρχει αυτή η τεχνολογία και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Αυτό μου θυμίζει Κάτι που είχε πει ο τελευταίος Γερμανός Κάιζερ πριν από 100 χρόνια. Είπε ότι το αυτοκίνητο είναι μια παροδική ε, μόδα ε, και ε, το άλογο θα δικαιωθεί τελικά. Ναι, δικαιώθηκαν οι ήπιοι στα αυτοκίνητα. ψηφιοποίηση έχουμε στην ε, τεχνολογία και στα μηχανήματα και τα μηχανήματα τα γεωργικά δεν είναι κάτι το παραδικό που θα χαθεί καθόλου. Θα ε, γίνει μηχανοκίνητη και η γεωργία, αυτό δεν δείχνει προς Το θέμα είναι τι επιπτώσεις θα έχει στη γεωργία και σε διάφορες μορφές γεωργίας. Αυτή είναι η ουσιαστική και σημαντική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Έγινε λόγος για τις μικρές επιχειρήσεις και τις εκμεταλλεύσεις σε δύσκολες περιοχές, ε, λιγότερο ευνοημένες και μειονεκτούσεις που είναι δύσκολο να χρησιμοποιείς μηχανήματα, αυτή η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο ε, τις ευνοημένες περιφέρειες, αλλά και άλλες περιφέρειες που είναι πιο δύσκολες. Για να μην χάσουν το τρένο, ε, ακόμα περισσότερα από όσα έχουν χάσει ήδη απέναντι στις πιο ευνοημένες περιφέρειες. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Τι γίνεται με τη συνεργασία ε, όπου οργανώνονται οι αγρότες για να ε, μοιράζονται τα μηχανήματα, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να έχει ε, δικά του μηχανήματα. Και στην Γερμανία και στην Αυστρία λειτουργούν καταπληκτικά αυτές οι δομές. Τώρα, Διαφωνώ με τον κύριο Χόσλινγκ. Ότι δεν είναι ελκυστικό για τους νέους αυτό. Φυσικά μπορεί να είναι ελκυστικό για 90-95% ε, των νέων αγροτών. Μπορεί κάποιοι να μην ενδιαφέρονται, αλλά οι νέοι αγρότες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ψηφιακά συστήματα, για τις έξυπνες μηχανές. Δεν έχω δει εγώ νέους που να μην θέλουν ε, να ε, εργάζονται με ε, υπολογιστές και έξυπνες συσκευές και μηχανήματα. Το αντίθετο. Δεν σας περιορίζω στο χρόνο αγόρευσης, αλλά παρακαλώ δείξτε και μια αυτοσυγκράτηση. Ο κύριος Νίκολσον. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία και η επιστήμη ε, μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στο μέλλον της Γεωργίας ε, και μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαδραματίσει και τέτοιο ρόλο. Μία από τις δυσκολίες που διαβλέπω εγώ σήμερα, αν ε, συζητά κανείς για μια οικογενειακή εκμετάλλευση, είναι το κόστος αυτής της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αν δείτε το κόστος ενός τρακτέρ σε σχέση με 30-40 χρόνια πριν, κάποιο γεωργός μου έλεγε ότι όταν αγόρασε το πρώτο τρακτέρ του, είπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό σήμερα, ε, γιατί του στήχησε δύο δεκάρες. Ε, κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι Γεωργοί. Δεν υπάρχει λόγος όμως να βλέπουμε στο παρελθόν και να θεωρούμε ότι τότε ήταν όλα ρόδινα. Ε, θα ξαναγυρίσουμε τι στις ε, άμαξες ε, στο κάρο με τα λογά. Θα πρέπει να δεχτούμε τις νέες τεχνολογίες, πρέπει να τις, να τις δεχτούμε. Το είπε και ο κύριος Τόρφον. έρχεται, υπάρχει αυτή η τεχνολογία και θα βελτιώνεται όσο προχωράμε. αν είναι κάποιο 55-60 ετών, δεν θα εναγκαλίσει φυσικά αυτέ τι τεχνολογίε, αλλά αν είσαι 25 και θέλει να εργαστεί το υπόλοιπο τη ζωή σου στη Γεωργία, σίγουρα θα τι αποδεχτεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούμε την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να ενθαρρύνουμε ενεργά τους πολίτες, τους γεωργούς ε, να το κάνουν αυτό. Ε, υπάρχει ορίζοντας 2020 και γι' αυτό το λόγο υπάρχει, για να γίνονται κάποια από αυτά τα πράγματα. Και πηγαίνουν πολύ πέραν των γνώσεων και της δικής μου της εμπειρίας όλα αυτά. Ζούμε σε καιρούς που πολύ δύσκολα μπορούμε να πείσουμε τους νέους ανθρώπους, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην εκμετάλλευση και εργάζονται εκεί. Αν θέλει κάποιος όμως να γίνει γεωργός, ε, η δουλειά είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα ε, και Πάσχα. Κάθε μέρα πρέπει να εργάζεσαι. Δεν μπορείς να πεις ε, στο γουρούνιο να, να φάει μόνο του την Κυριακή. πρέπει λοιπόν να κάνουν ε, αυτή τη δουλειά. Βλέπουν τους φίλους τους την Παρασκευή το απόγευμα να σταματάνε τη δουλειά και να ξανάρχονται τη Δευτέρα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πείσουμε κάποιους ανθρώπους να μείνουν στην εκμετάλλευση και να κάνουν κάποιες από τις εργασίες. Δεν ξέρω και η συνάδελφος εδώ να αναφερθεί ε, ε, ίσως το θέμα όταν θα μιλήσει είναι αυτά που βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, υπάρχει εξάρτηση από τους μετανάστες που πρέπει να έρθουν να κάνουν κάποιες από τι εργασίες που κανείς δεν θέλει να κάνει στην εκμετάλλευση. Είτε λοιπόν θα δεχτούμε τεχνολογία για να κάνει αυτές τις δουλειές ή θα προσλάβουμε ανθρώπινο δυναμικό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, μα δώσετε κάποιες ιδέες. Ε, Στη σελίδα 27 της μελέτης σας λέτε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Γεωργία να εξαρτάται από μη γεωργική παραγωγή για τεχνολογία και για μηχανήματα μη ευρωπαϊκή παραγωγή για τεχνολογία και μηχανήματα για αυτή τη μορφή στη γεωργία ακριβία. Γιατί αυτό, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από τον ορίζοντα 2020 ή άλλα τεχνολο... Ε, κονδύλια για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή τεχνολογία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια πρόταση. Θα πρέπει να αναθέσουμε σε κάποιο ουδέτερο, αμερόληπτο, μια, την εκμόνηση μελέτης ε, που θα προσπαθεί να βρει πόσο καιρό ξοδεύουμε για να ε, συζητούμε για τις τράπεζες, τους μεγάλους παραγωγούς μηχανών που κάνουν το βίο αβίωτο και ψήνουν το ψάρι στα χείλη των γεωργών. Πόσες χρόνο αφιερώνουμε να συζητούμε για αυτούς. Επίσης, τι επενδύσεις θα χρειαζόταν μία εκμετάλλευση για να κρατήσει δύο μονάδες εργασίας ε, στην ε, γεωργία, σε τέτοιου είδου γεωργία ακριβίας. Δεύτερον, τι αντίκτυπο θα έχει μια τέτοια επένδυση σε ό,τι αφορά τη χρέωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τρίτον, τι επίπεδο τιμών θα πρέπει να εφάρμοζε ο Γιώργος για να, είναι, για να αποσβέσει τις επενδύσεις του, για να είναι συμφέρουσες. Γιατί μιλούμε για επενδύσεις, αλλά η πραγματικότητα των Γιωργών, ανδρών και γυναικών ε, είναι διαφορετική, γιατί οι τιμές των προϊόντων είναι πολύ χαμηλές. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Έγινε κάποιος, ε, κάποια μελέτη αντικτύπου για το πώς θα επηρεάσει τέτοιου είδους ε, γεωργία, γεωργία ακριβία στη συγκέντρωση της παραγωγής σε μεγάλες μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες ε, από τον καλεσμένο μας. Δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις απορίες μας. Μερικά ερωτήματα θα πρέπει μόνοι μας να τα απαντήσουμε, να τα αφήσουμε για άλλη φορά. Κύριε Μακιντάιρ. Εγώ είμαι. Καταρχήν, συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή της παρουσίαση. γιατί πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ αυτό το θέμα και ω μέλο του πάλι του ΣΤΟΑ παρακολουθώ αυτό το ζήτημα και γνωρίζω την πρόοδο που έγινε και τη μελέτη αυτή για τη γεωργία ακριβία. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου και να εξάρω και εγώ την σημασία, τη σπουδαιότητα που έχει η Γεωργία Κρυβίες και τη σημασία που έχει η οθέτηση τέτοιων τεχνικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την τύχη να είμαι εισηγήτρια της Επιτροπής Γεωργίας στην έκθεση για τις τεχνολογικές λύσεις για μια αηφόρο γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το επίθετο αηφόρος είναι πολύ σημαντικό στον τίτλο της έκθεσης, γιατί το θέμα είναι η τεχνολογία να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε μια πιο αηφόρο γεωργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα West Midlands, στη δική μου περιφέρεια, έχουμε ένα πανεπιστήμιο ε, και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι έχουν επισκεφτεί μαζί μου αυτό το πανεπιστήμιο που πραγματικά έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες και πολύ σημαντικές εργασίες στον τομέα αυτό. Να σας πω λοιπόν ε, ποιες είναι κάποιες ε, προσπάθειες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το 2011 το πανεπιστήμιο αυτό έχει ε, εισάγει ένα σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας ε, στην Γεωργία, το Πανεπιστήμιο Harper Adams, και ε, τα μηχανήματα θα μπορούν να, να, έχουν, να επεξεργάζονται 86% μιας αρρώσιμης καλλιέργειας και 56% των ε, ε, βοσκοτόπων. Φυσικά είναι τεράστια η βλάβη από τη συμπίκνωση του εδάφους που, που είναι αποτέλεσμα αυτών των, των μηχανημάτων. Και γι' αυτό με το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας στη Γεωργία θα μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Άλλωστε υπάρχουν τεχνολογίες και μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά με την ανάπτυξη ενός ε, ε, διαφορετικών μορφών τεχνολογίας μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο της ε, συμπίκνωσης του εδάφους. Επίσης, μπορούμε να, να εξολοθρεύσουμε τα ζυζάνια με τη χρήση λέιζερ, όχι με ζυζανιοκτώνα κατά ανάγκη. Γιατί να μην σκοτώνουμε τα ζυζάνια με, με λέιζερ. Ακόμη και η βιολογική παραγωγή είναι υπέρ αυτής της μεθόδου. Επίσης, αν χρησιμοποιήσουμε μη παντρωμένα ε, αεροσκάφη δεύτερης γενιάς, τα drones, μπορούμε να ε, βγάλουμε φωτογραφίες που θα είναι πολύ χρήσιμες για τη γεωργία ακριβίας. Υπάρχει τεράστιο πεδίο πρόοδου λοιπόν. Δεν χρειάζεται να περιοριστούμε κατά ανάγκη στα τεράστια μηχανήματα, στον κόδι μηχανήματα που είναι και πολύ δαπανηρά και που ούτως ή άλλως η ανάπτυξή τους είναι πολύ χρονοβόρα. Και αλλά το κόστος πιστεύω ότι δεν θα ε, είναι κατά ανάγκη αστρονομικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που μας είπε ο κύριος Νίκολσον, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επικεντρωθούμε σε εφαρμοστική έρευνα, όχι μόνο ε, θεωρητική, σε εφαρμοσμένη έρευνα για να ε, μετατρέψουμε τις ιδέες σε έμπρεκτες λύσεις, να τους δώσουμε σάρκα και οστά για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητά τους από τους γεωργούς. Και τότε θα δούμε τους καρπούς και φυσικά ανα... εμπλέκοντας τους γεωργούς σε αυτή την εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν ξέρω αν ήταν καλή η απόφαση μου να μην σας περιορίζω στο χρόνο αγόρευσης. Κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ. Ως μέλος του πάρελ του ΣΤΟΑ. Θα ήθελα φυσικά να χαιρετήσω ε, και να επενέσω το ερευνητικό έργο ε, του πάνελ και πιστεύω ότι οι χρήσιμες αυτές τις παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη και στην λήψη κάποιων πολιτικών αποφάσεων και ευελπιστώ να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε κάνει ένα υπολογισμό για το πως η μέση γεωργική εκμετάλλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει προκειμένου να εξοπλιστεί με τις απαραίτητες τεχνολογίες ε, για να ασκήσει τέτοιου είδους γεωργία, γεωργία ακριβίας. Μας υπενθυμίσατε την, ε, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γεωργικών κοινοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επενδύσουμε στην κατάρτιση των γεωργών και στι νέες τεχνολογίες που είναι απαιτητικέ και περίπλοκες, ιδιαίτερα για του πιο ηλικιωμένου γεωργού. Επίσης, ε, θα ήθελα να ε, κατατοπίσετε, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, αμφιβολίες και να μου πείτε τι ακριβώς εννοούμε με την ε, γεωργία ακριβίας μιλούμε μόνο για τη χρήση τεχνολογίας, ρομπότ, δορυφόρων και άλλων τεχνολογικών επιτεγμάτων για την άσκηση των γεωρικών δραστηριοτήτων. Ή περιλαμβάνει η γεωργία ακριβίας, όπως ακούμε μερικές φορές, και την ε, γενετική τροποποίηση και τη χρήση γενετικών μεθόδων. Γιατί αν μιλούμε για το δεύτερο που ανέφερα, τη γενετική τροποποίηση, δεν συμφωνώ με τέτοιου είδου γεωργία ακριβία, γιατί θεωρώ ότι στην Ευρώπη δεν χρειαζόμαστε γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. Έχουμε και αρκετέ γνώσει και αρκετού πόρου για να παράγουμε και να αυξήσουμε την παραγωγή μα με ε, φυσικό τρόπο που θα σέβεται και το περιβάλλον και τη φύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ, που είναι ο τελευταίος, που επειδή καθυστέρησε, τον τιμωρώ και του δίνω μόνο ένα λεπτό γιατί ήταν απόν σε μεγάλο τμήμα των εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι ξέρουν τις απόψεις μου και η γεωργία χρειάζεται τις επιστημονικές εξελίξεις και τις τεχνολογικές και το θέμα δεν είναι το θέλουμε εμείς ή όχι, είναι τι πολιτικές αποφάσεις θα πάρουμε, γιατί θα επέλθουν αυτές οι αλλαγές. Λέτε ότι τα λεφτά θα τα φάνε οι μεγάλοι όμιλοι που παράγουν τα γεωργικά μηχανήματα. Κοιτάξτε. Έχει τύχει να χρειαστεί να αρμέξω όταν ήμουν νέο, ήμουν κακόκεφο και αγελάδα κακό και φύγε ευτυχώ που έχουμε τώρα μεκτικέ μηχανέ και είναι και για του δύο καλύτερα. Ε, το πρόβλημα ποιο είναι. Η προστασία των δεδομένων λέτε. Περίεργο δεν είναι αυτό και άλλοι συνάδελφοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν να το λύσουμε. Γιατί έχουμε σε λίγο το έξυπνο ψυγείο ε, που θα διαχειρίζεται το τι θα φας γιατί πάχινες. Ε, τα δεδομένα αλλάζουν και αλλάζει και η διαχείρισή τους. Η προστασία των δεδομένων είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί τελικά η αξία των δεδομένων θα υπερβεί την αξία του μηχανήματος, έτσι. Ε, δηλαδή, εμείς θα πρέπει να διαμορφώσουμε έτσι την πολιτική μας για να το ρυθμίσουμε αυτό. Και το δεύτερο που με απασχολεί και με βασανίζει στην γεωργία ακριβία είναι ορισμένα εχθρικά ε, πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί και θέλω να με βοηθήσετε. Αν είναι τόσο περιορισμένο και οι εταιρείε κάνουν και τη διαφήμισή τους με τεράστια τρακτέρ, ε, τεράστια χωράφια, φεύγεις το πρωί και όταν για επιστρέψεις είναι μεσημέρι, χρειάζεται και μια αποδοχή από την κοινωνία. Η γεωργία ακριβίας είναι για τη βιομηχανική ε, γεωργία. Αν κάτι τέτοιο πιστέψει η κοινωνία, χάσαμε το παιχνίδι και την αποδοχή. Θα πρέπει λοιπόν η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος να είναι προς όφελος όλων. Έχετε συμβουλές πού μπορούμε εμείς να το ε, προβάλλουμε να το προωθήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ πολύ έξυπνα ε, με, ε, μου μίλησε μιλώντας για, αυτές τις, για, για αυτά τα έξυπνα ψυγεία. Εμένα σκεφτόταν όταν ανέφερα αυτό το παράδειγμα. I Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και για τις παρατηρήσεις. Ε, πιστεύω ότι ε, με διαφορετικούς τρόπους ε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες ερωτήσεις και πιστεύω ότι οι περισσότερες από αυτές απαιτούν μια μακροσκελή μελέτη ή μια μακροσκελή απάντηση για τους μικρούς γεωργούς. Την άλλη φορά, λέει ο Πρόεδρος, υπάρχει μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τους ναι, μικρούς γεωργούς. Ε, εγώ να σας κάνω την άλλη ερώτηση. Αν κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν, θα έχουμε μια γεωργία η οποία στα δεκα, ε, επόμενα 15-20 χρόνια πώς θα είναι. Αν κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και δεν ενθαρρύνουμε ε, κάποιου ε, να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι οι νέοι γεωργοί που συνάντησα εγώ και μεταξύ φίλων αλλά και στι διάφορες χώρες ε, είναι ενθουσιώδης ε, εάν ε, τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια εκμετάλλευση που έχει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες. Και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι απλώς ε, ογκώδη μηχανήματα. Η τεχνολογία είναι ένας πολύ ευρύς όρος, ε, τον οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου γενικώς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εάν ένας γεωργός έχει ένα έξυπνο τηλέφωνο, καλύτερο από το δικό μου, και όταν πηγαίνει στο χωράφι του βγάζει φωτογραφίες. Μπορεί να είναι ένα μικρό χωράφι. Και οι φωτογραφίες αυτές περνούν από το υπολογιστικό νέφος και λαμβάνει μια απάντηση ότι εδώ, σε αυτή την περιοχή, υπάρχει ε, ασθένεια και εδώ σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει. Ή εκεί υπάρχει έλλειψη αζότου και εκεί υπάρχει ε, υπερβολική παρουσία αζότου. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη εκμετάλλευση, μπορεί κάλλιστα να το κάνει αυτό και ήδη μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει. Χρησιμοποιεί λοιπόν τεχνολογία και γνώσεις οι οποίες παράγονται κάπου. Διότι εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι απλώς ε, ε κοιτώντας με τα μάτια του μπορεί να ε, καταλήξει σε αυτές τις ερμηνείες. Μπορεί να φταίω εγώ όμως. Εγώ όταν εργαζόμουν στην εκμετάλλευση του πατέρα μου δεν μπορούσα να το καταλάβω, το ένστικτό μου δεν με βοηθούσε πάντα και πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Ε, γι' αυτό χρειάστηκε να πάω και στο πανεπιστήμιο. Τον βοηθά λοιπόν. Όταν λέμε ε, να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα, είναι ένας τρόπος να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε παραγωγή η οποία θα είναι περισσότερο στραμμένη στην αγορά, να έχουμε πληροφορίες για το τι θέλει η αγορά και ε, να χρειάζεται ίσως λιγότερη προσπάθεια ή με τα ίδια να, κάνουμε, να καταλήγουμε σε καλύτερο εισόδημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στο μέλλον να ξέρουμε τι θέλει η αγορά. Και ποιο βρίσκεται πίσω από αυτό. Όλοι βρισκόμαστε πίσω από αυτό. Η πρόσβαση στην αγορά θέλουμε να δίνεται μόνο σε ε, γεωργούς που εμπιστευόμαστε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είδαμε την κρίση στην Ευρώπη. Είδαμε τα σούπερ μάρκετ, τους λιανοπολιτές, αλλά νομίζω ότι όλοι στην αλυσίδα θέλουν να είναι βέβαιοι ότι αυτό που αγοράζουν είναι αποδεκτής ποιότητας και ε, ασφαλές. Και ε, ούτως ή άλλως το μεγάλο παιχνίδι είναι η καταγραφή όλων αυτών και υπάρχουν ε, και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία εισήχθησαν και γνωρίζουν οι Γεωργοί ότι πρέπει πλέον να κάνουν αυτό που λένε και να καταγράφονται όλα αυτά κάπου και αυτό φυσικά είναι δαπανηρό. Πρέπει να πληρώνουμε περισσότερα. Νομίζω ότι αρχικά ε, αυτοί που αγόραζαν λιανική ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο, αλλά δεν αρκούσε αυτό στη συνέχεια. Ήταν ε, ο τρόπος που λειτουργεί η ζωή νομίζω. Και αυτή η νέα τεχνολογία, η καταγραφή είναι πολύ εύκολη διότι σκανάρετε τον κώδικα του προϊόντος και ξέρουμε τι ε, ε, έχει αυτό το προϊόν. Ε, και νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι όταν πηγαίνουμε στο κατάστημα, εγώ κάνω και επίδειξη ορισμένε φορές, δεν είμαι πολύ καλός. Κάποιο όμω πρέπει να μα δώσει αυτά τα δεδομένα, πρέπει να παράξει αυτέ τι πληροφορίε. και το τι έκανε το καταγράφει ο γεωργός και γίνεται είτε στη βιολογική γεωργία είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή γεωργία. Αυτό είναι αυτό που θα του ζητάμε, διότι ζητάμε και ε, ε, από τους ε, βιολογικούς καλλιεργητές τι έκαναν. Και περιμένουμε διαφορετικές απαντήσεις. Και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Στη βιολογική καλλιέργεια περιμένουμε να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα του εδάφους κλπ. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε και τους γεωργούς. Είναι ακόμα στα σπάργανα αυτό, αλλά θα έρθει στη συνέχεια. Ε, να ενημερώνουμε τους γεωργούς για τη βιολογική ποιότητα του εδάφους, γιατί αυτό έχει σημασία και για την διάρθρωση του εδάφους και τη διάβρωση του εδάφους, προκειμένου να αποφύγουμε διάβρωση η τεχνολογία αυτή θα είναι διαθέσιμη και σε άλλους ε, γεωργούς και όταν έχουμε περιτροπής καλλιέργειες ε, γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος ε, για να διαγείρουμε την μικροβιακή ζωή του εδάφους και η μικροβιακή ζωή του εδάφους είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη φυτοϊγεία και για την αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών. κατέγραψα και κάποιες ε, ερωτήσεις εδώ για ίδια χρήση. Τώρα, η χρήση και η ιδιοκτησία των δεδομένων είναι πολύ σημαντικό θέμα που αποσχολεί και πανεπιστημιακές κοινότητες και εσάς φαντάζομαι. Ε, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. από κάποιες ε, εταιρείες που έχουν προκύψει από τα πανεπιστήμια που χειρίζονται τα δεδομένα. Όταν ο Γιώργος δεν θέλει να δώσει τα στοιχεία, ε, δεν μπορεί φυσικά να ε, λάβει και πληροφορίες από τις γνώσεις προς αποκύπτουν από τα δεδομένα. Το να έχει κάποιος αν του ε, γεμάτο δεδομένα και κλειδωμένο ε, δεν το κάνει σίγουρα πιο έξυπνο. Εάν μπορεί κάποιος να επεξεργάζεται τα δεδομένα θα αποκομίσει κέρδος από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτός που παρέχει την υπηρεσία και κάνει την ανάλυση θα είναι αυτός ο οποίος θα υποφελείται. Δεν το πιστεύω αυτό, πιστεύω ότι και ο Γιωργός θα υποφελείται. Πώς μπορούμε να ασφαλίσουμε ότι θα τηρείται η εμπιστευτικότητα. Αυτή είναι μια συζήτηση που χρειάζεται άλλες δύο μέρε κύριε Πρόεδρε. Τα γνωρίζουμε όμως όλα αυτά και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της ψηφιοποίησης όλης της κοινωνίας. εγώ έχω ηλιακά πάνελ, η εταιρεία που τα εγκατέστησε φαίνεται να γνωρίζει όλες αυτές τις πληροφορίε για τα πάνελ που έχω. Ε, τουλάχιστον εγώ θα μπορώ να παρέμβω βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να τα δω αυτό στα φωτοβολταϊκά πάνελ. Κάτι αντίστοιχα υπάρχει. Τώρα, ψηφιοποίηση σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό είναι θέμα τεχνολογίας. Αν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών θέλουν να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες εκεί. Τουλάχιστον όμως υπάρχει πρόσβαση στις περιοχές αυτές. Είναι ε, πολλές οι γνώσεις αυτές για τους νέους ανθρώπους και νομίζω ότι αν υπάρχει καλύτερη παιδεία που θα λάβει υπόψη της και την γεωργία ακριβίας, θα μάθουν τα παιδιά να εργάζονται με τα έξυπνα τηλέφωνά τους και με την αποτελεσματική τεχνολογία και θα μάθουν ότι θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν αυτό στην εκμετάλλευσή τους. Ή θα μπορούν να συμβουλευτούν βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, θα μπορούν να συμβουλευτούν ε, πληροφορίες ε, για διάφορους ε, γονότυπους που πρέπει να λάβουν υπόψη στα φυτά και μάλιστα η Γεωργία Κρυβίας προσπαθεί να βελτιστοποιήσει το συνδυασμό ε, του περιβάλλοντος, του εδάφους δηλαδή και του γονότυπου και ε, την τεχνολογία. Δεν έχει καμία σχέση με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Αλλά επειδή υπάρχει αραβόσιτος και χρησιμοποιείται ε, και υπάρχουν και ζυζάνια που αναπτύσσουν ρίζες οι οποίες πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα ε, βαθιά στο έδαφος. Θα είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν η καλλιέργεια σε ξηρέ περιοχές σε σχέση με άλλες μορφές. Αυτά είναι πολύ καλά να τα γνωρίζει και να τα χρησιμοποιεί ο Γιώργος, να έχει πρόσβαση σε αυτές τις προφορίες και να μπορεί να γνωρίζει την περιεκτικότητα σε υγρασία του εδάφους ε, και να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη καλλιέργεια. Και φυσικά Νομίζω ότι και οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πληροφορίες ε, για το έδαφος και το γονότυπο για να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τη σύσταση των υδάτων που έχουν στο έδαφος. Τώρα, συνεργασία και εξειδίκευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει στη γεωργική κοινότητα. Πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το μέλλον θα δείξει. Ε, θα τα ξαναδούμε αυτά σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια για να δούμε τι συνέβη. Νομίζω ότι όσον αφορά τις γεωργικές κοινότητε θα υπάρχει εξειδίκευση ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ε, μικροί γεωργοί μπορεί να, μείνουν, να παραμείνουν μικροί γεωργοί, αλλά θα είναι απόλυτα εξειδικευμένοι. Και γιατί ένας γεωργός να ξέρει τα πάντα για ό,τι συμβαίνει στην εκμετάλλευσή του, διότι αν ζει σε μια γεωργική κοινότητα, οι συνεταιρισμοί θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν ιδιαίτερα θα μπορεί να μοιράζεται εξοπλισμό, αλλά και γνώσεις και πυρογνωμοσύνη. Και αυτό φυσικά διδάσκεται. Ιδίω αν ανανεώσουμε και τα εκπαιδευτικά συστήματά μας. Αν με ρωτήσετε τι χρειάζεται να επενδύσει ε, μια εκμετάλλευση για να αρχίσει μια γεωργία ακριβίας, Μπορεί να είναι ελάχιστη επένδυση, μια προσαρμογή απλή της δόσης ε, των φαρμάκων και των λιπασμάτων ανάλογα με στοιχεία και δεδομένα που ε, μεταφέρει και διαβιβάζει με το τηλέφωνο του. Και αυτό είναι, Γεωργία ή να ψεκάζει τα λοιπάσματα πιο κοντά ε, στα ριζικά συστήματα των φυτών για να απορροφούν καλύτερα και όχι γενικά να ραντίζει όλο το χωράφι. Ναι, Πρόεδρε, ε, δεν έχω χρόνο μάλιστα. Αυτά. Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω ώρες για τη Γεωργία, όπως ε, όλοι εδώ άλλωστε. Ελπίζω να απάντησα περισσότερες ερωτήσεις σας. Αν έχετε περισσότερες ακόμα, μέσω του πάνελ στο ή με το προσωπικό μου email μπορείτε να με ρωτήσετε και με χαρά να απαντήσω. Και πάντα τα συζητάμε όλα. Γιατί ό,τι πω δεν σημαίνει ότι είναι πάντα απόλυτη αλήθεια. Εμεί προσπαθούμε να λέμε την αλήθεια, αλλά μπορεί να μας έχουν διαφύγει και κάποια θέματα από τη συζήτηση γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Και ο καθηγητής Ντεκάστρο ε, επιβεβαίωσε ότι είχαμε σήμερα την πολυτέλεια για μια πιο ακαδημαϊκή συζήτηση, χωρίς δηλαδή περιορισμό χρόνου. Συμβαίνει και αυτό που και που. Σπάνια όμως. Πάντως, σίγουρα αυτές οι έλεγες ξεκίνησαν, δεν μπορούμε να τις συγκρατήσουμε. Ίσως θα μπορούσαμε όμως να τις κατευθύνουμε. Λαμβάνοντας, ε, λαμβάνοντας υπόψη και στη μεταρρυθμίση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω ότι τις παρατηρήσεις και τα πορίσματά σας θα τα αξιοποιήσουμε στο μέλλον κατά τη συζήτηση και διαμόρφωση της μελλοντικής κοινή γεωργικής πολιτικής. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξής μας, τις ε, γενικές διατάξεις ελέγχου των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συντονιστές ε, έλαβαν την απόφαση ε, να συντάξουν γνωμοδότηση επί της, επί της ε, έκθεσης της ε, Επιτροπής Ομικών Υποθέσεων για την Επιτροπολογία. Ο κύριος Άγερ είναι ο εισηγητής έκθεσης, ενώ συντάκτης της δικής μας γνωμοδότησης είναι ο κύριος Ροπέ. Ο κύριος Ροπέ θα λάβει τώρα το λόγο για να σε ενημερώσει για τις γενικέ αρχέ και του κανόνε σχετικά με του τρόπου ελέγχου τη άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησής μου για την επιτροπολογία. Η αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή που θα εκπονήσει και έκθεση είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, εμείς όμως αποφασίσαμε να καταρτήσουμε γνωμοδότηση για τις προτάσεις και τα προβλήματα της επιτροπολογίας που αφορούν και την ΚΑΠ και την ε, ε, Γενική Διαδικαστική Οργάνωση. Η διαδικασία της επιτροπολογίας ε, δίνει την ευκαιρία στους εθνικούς εμπειρογνώμονες να εξετάσουν όλες τις ε, ευρωπαϊκ... όλα τα ευρωπαϊκά νομοθετικά ζητήματα και για αυτό το λόγο η συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και των ε, αρμοδίων τμήματων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, θεσπίζουν δευτερογενές ε, ενωσιακό δίκαιο μέσω των εφαρμοστικών και κατεξοδότηση πράξεων και αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Πολύ συχνά οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αποφεύγουν να εκφέρουν γνώμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει εκείνη την ευθύνη και προβαίνει σε αποφάσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση των κατεξοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί απλώ να τι εγκρίνει ή να τι απορρίψει. Δεν έχει όμω το δικαίωμα να τι τροποποιήσει. Ω εκ τούτου πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την δημοκρατική νομοποίηση της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων μέσω της επιτροπολογίας και να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διαβούλευσης προκειμένου να γίνουν πιο υπόλογα τα κράτη-μέλη. Επίσης, σημαντικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να επαφίονται σε ένα μικρό αριθμό χωρών μελών. Κάτι τέτοιο θα ισχύσει αν δεν καταμετρώνται οι αποχές στη λήψη των αποφάσεων, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω λοιπόν να προτείνουμε στην γνωμοδότησή μας το εξή. Καταρχήν η αρχή της προφύλαξης, μεγαλύτερη λογοδοσία των κρατών μελών και ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας καθώς και αποτελεσματική έλεγχη της εντολής ε, που χορηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ακράδοντα ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε ευρέω την αρχή της προφύλαξης, ώστε οι άδειε για τη χρήση υλικών ε, και προϊόντων να χορηγούνται μόνο μετά από απόφαση ε, που έχει ληφθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή. Και αυτό κυρίως ισχύει για θέματα που αφορούν την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος ή την υγεία φυτών, ζώων, ανθρώπων, καθώς και την ασφάλειά τους. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας επιτροπολογίας. Γι' αυτό προτείνω να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για να φαίνονται οι θέσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών και το πώς ψήφισαν και να αιτιολογούνται και οι απόψεις τους. Επίσης προτείνω να δημοσιεύονται οι πληροφορίες για τη σύνθεση των επιτροπών και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις καθώς και πληροφορίες για τις αρχές που εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Επιτροπή Προσφυγών δεν ε, εξυπηρετεί σε τίποτα, γιατί τα αποτελέσματα ψηφοφορία ψηφοφορίας Επιτροπή προσφυγή Προσφυγής ταυτίζονται πλήρω με τα αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας ψηφοφορίας. Γι' αυτό προτείνω να καταργηθεί η Επιτροπή Προσφυγών. Είναι τελείως απέριτη και άχρηστη. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν την εφαρμοστική εντολή που ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ανακαλέσουν την νομοθεσία ανα πάσα στιγμή. Αυτό είναι το περιεχόμενο της γραμμοδότησης που υποβάλλω στην Επιτροπή Γεωργίας και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια ε, τις παρατηρήσεις και τις επικρίσεις και προσβλέπω σε συνεχή και αγαστή συνεργασία και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Ροπέ. Πολύ αυτές οι προτάσεις σας. Περνάμε στη συζήτηση. Η κυρία Γκέρλινγκ ζήτησε πρώτα το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους στόχους του εισηγητή όπως του παρουσιάζει στην έκθεσή του. Έχει απολύτως δίκιο. Είναι υπόλογα τα κράτη-μέλη και να λογοδοτούν όταν παίρνουν αυτές τις αποφάσεις μόνιμες επιτροπές. Είναι απολύτως σωστό να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά το παρακάνει για τη διαφάνεια, πιστεύω, ο εισηγητής. Δηλαδή να έχουμε δημόσια πλήρη έκθεση και αναφορά ε, το πόσα κράτη ψήφισαν και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Αλλά αυτό που ζητάει, συγγνώμη το παραφράζω λίγο, αυτό που ζητάει είναι πλήρη αιτιολόγηση ε, του τρόπου με τον οποίο ψήφισαν τα κράτη-μέλη νομίζω είναι υπερβολικό. Και θα ε, γνωρίσει φοδρές αντιστάσεις και ο Μέσδηλος ε, ως απάντηση. Τώρα ζητάμε πλήρη δικαιολόγηση από τα κράτη-μέλη, το πώς ψήφισαν για κάθε νομοθέτημα έτσι, παραγόγου δικαίου. Ε, είναι υπερβολικό και μπορεί να πάρουν αποφάσεις ε, λόγω αυτού που δεν θα έπαιρνε. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, αλλά όχι αυτά τα υπερβολικά. Ο εισηγητής μας σε όλη την έκθεση θεωρεί ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε οι εκπρόσωποι των μικρών κρατών μελών, δηλαδή να μην λαμβάνονται αποφάσεις από μια χούφτα μεγάλες χώρες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ελεύθερη βούληση και τα υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που παίρνουν μια απόφαση να μην ψηφίσουν. Όπως και εμείς ε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καμιά φορά απέχουμε. Ή καμιά φορά δεν ψηφίζουμε γιατί βαριόμαστε και δεν σηκώνουμε χέρι ή δεν έχουμε άποψη ή δεν θεωρούμε ότι έχουμε αρκετή πληροφόρηση για να εκφράσουμε μια άποψη. Η αποχή καμιά φορά μπορεί να είναι πάρα πολύ λογική στάση. Αλλά δέχομαι ότι η αποχή ε, σε μόνιμες επιτροπές ε, έχει προσλάβει πλέον μια πολιτική χρειά. Ε, σε πολλές επιτροπές δίδουν οδηγίες στα κράτη-μέλη στους εμπειρογνώμονες να μην ψηφίσουν ακριβώς για να αποφύγουν να είναι τμήμα της απόφασης. Όταν ληφθεί απόφαση, εάν ληφθεί τέτοια απόφαση, καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι δική μας δουλειά να προστατεύουμε αυτά τα κράτη-μέλη. Και για ποιο λόγο να χρήσουμε τους εαυτούς μας προστάτες των μικρών χωρών μελών. Καμιά φορά δεν ψηφίσουν και μεγάλες χώρες και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο στρεβλωτικό. Ας πούμε αν έχει τη Γερμανία, την Ισπανία, το Μένο Βασίλειο να μην ψηφίσει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ χειρότερο σε σχέση με πολλά μικρά κράτη-μέλη. Αν ένα κράτος επιλέξει να πει στους εμπειρογνώμονες να μην ψηφίσουν, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση λοιπόν συχνά σε μια επιτροπή επιρρογνωμόνων που κατά βάση δεν θα πρέπει να είναι πολιτική εντό εισαγωγικών, θα πρέπει να βασίζεται ε, στην γνώμη των επιρρογνωμόνων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αποφασίζουν τα κράτη-μέλη επιρρογνώμονε να μην ψηφίσουν, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή αυτή η απόφαση. Υπάρχει διαδικασία των προσφυγών. Ε, αν ε, έχει το ίδιο αποτέλεσμα εκεί, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να απέχει ε, στο πρωτοβάθμιο ας πούμε όργανο και δεν θέλει να, να προχωρήσει, να συμμετέχει στις προσφυγές, νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ λογική ε, απόφαση. Δεν συμφωνεί ο εισηγητής. Αν δεν υπάρχει ειδική ε, πλειοψηφία ε, στην αρχή μειώνεται το σύνολο των ανθρώπων που μπορούν να ψηφίσουν σε δεύτερο στάδιο στην προσφυγή και αυτοί θα πρέπει να είναι εκείνοι που επέλεξαν να ψηφίσουν και που έχουν γνώμη, όχι όλοι. Και είναι και ένας κομψός τρόπος ε, και εύσχημος να βγούμε από αυτό το ε, αδιέξοδο που έχουμε καταλήξει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ βαθιστόχαστες αυτές οι παρατηρήσεις και πολύ εύστοχες και ουσιαστικές. Ο κύριος Ντενανό. Ναι κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα του έργου του. Ε, είναι άχαρο το θέμα, ε, νομικό, τεχνικό, αλλά και πολύ πολιτικό. Η επιτροπολογία είναι πολύ σημαντική για την ε, εφαρμογή βασικών κειμένων που ε, αφορούν για τη γεωργία, ας πούμε, την κυκλοφορία στην αγορά φυτογενομικών προϊόντων ή ακόμα και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτά τα θέματα που είναι αρκετά περιπλοκά και οι στάσεις θα πρέπει να ε, τεκμερώνται από ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες και διαφανείς επιστημονικές θέσεις. Διάβασα το κείμενο για την αρχή της προφύλαξης. Ε, δεν είμαι καθόλου πεπισμένος αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και ο εισηγητής, ε, για το κατά πόσο θα λυθούν τα προβλήματα. Εκφράζω κάποιες αμφιβολίες Ε, συστηματικά ε, απορρίπτεται η ε, οποιαδήποτε έγκριση αδειοδότηση κυκλοφορίας προϊόντων στην αγορά όταν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία στην Επιτροπή Προσφυγών. Σίγουρα θα είναι πολλές οι διενέξεις και οι δικαστικές αντιπαραθέσεις. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια χωρίς όμως να εκτίθενται και να κατονομάζονται οι εμπειρογνώμονες και το πώς ψήφισαν στην κάθε ε, επιτροπή. Θα πρέπει ενδεχομένω και το Συμβούλιο να γνωμοδοτεί ε, για θέματα πολύ σημαντικά και πολιτικά με έντονες συζητήσεις και τεκμηριωμένες. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα. Ενδιαφέρον ο τρόπος ε, με τον οποίο βλέπει το θέμα και κατανοητός. Καλό που κάνουμε τη συζήτηση αυτή για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, αλλά εγώ βλέπω μια διαφορά ανάμεσα σε εκείνο που θέλει ε, ο εισηγητής ε, και αυτό που θέλει η δική μας πολιτική ομάδα. Ας προσπαθήσουμε να παραμένουμε όσο γίνεται περισσότερο στις επιστημονικές απόψεις, στις επιστημονικές επιτροπές. Ο εισηγητής τι λέει. με αυτό που προτείνει είναι πολύ απλουστευτική η πρόταση και θα καταψηφίζονται ε, ε, πολλά τέτοια φυτογειονομικά προϊόντα, ακόμα και ε, γενετικά τροποποιημένα, γιατί λέει αν δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία θα πρέπει συστηματικά να απορρίπτονται. Δεν θα πρέπει να πολιτικοποιούμε αυτό το θέμα όπως κάνουμε τώρα και να ψάξουμε να βρούμε μια λύση με λιγότερο πολιτικοποιημένο τρόπο και να εμπιστευόμαστε για να ακούμε περισσότερο τα επιστημονικά μας όργανα. Και να ακολουθήσουμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουν λόγο τα κράτη-μέλη εφόσον έχουν και σαφή άποψη και όχι να απέχεις και μετά να άρχισε να λες τη γνώμη σου. Τροπολογίες δεν θα κάνουμε, θα το συζητήσουμε στο εσωτερικό της ομάδας και βλέποντας και κάνοντας και είμαι πρόθυμος και προσβλέπω στη συνεργασία με τους άλλους και τους Ο κύριος Γιάρ, ευχαριστώ πολύ. Τρία σχόλια. ε, ως θύμα, γιατί καμιά φορά είμαστε θύματα της διαδικασίας στην Επιτροπή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προετοιμάζει, ε, το πρώτο, δεύτερο. Θυμάμαι τη τελευταία κατεξοδότηση πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτιάχνει κολοσσούς κατασκευάσματα νομοθετικά ε, γίγαντες. Καλό, είναι να έρχονται πιο μικρά νομοθετήματα και τέτοιες πράξεις για να μπορούμε να παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε διαφορετικά προβλήματα στην ίδια νομική πράξη, νομοθετική. Και τρίτον, στο Συμβούλιο υπάρχει κάτι που με ενοχλεί, οι αποχές. Διότι Εντάξει, δημοκρατία και τα λοιπά, όλα είναι νόμιμα και ορθά. Και στο κοινοβούλιο έχουμε αποχές στην ψηφοφορία, πλην όμως τα πράγματα δυσκολεύουν όταν χρειάζομαι μια ειδική πλειοψηφία, γιατί η αποχή de facto θεωρείται αρνητική ψήφος. Και ποιο σηκώνει αυτό το σταυρό, τα κράτη-μέλη που έχουν άποψη. Μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο τουλάχιστον οι αποχές να μην μετράνε ως αρνητικές και να επιβαρύνουν τη διαδικασία. Δεν λέω να αναγκάζουμε όλα τα κράτη-μέλη να ψηφίζουν, αλλά αν θέλουν να πούν όχι, ας πούν όχι, όχι μέχρι την αποχή να εμποδίζουν ε, την λήψη απόφαση. Δημοκρατία σημαίνει να είσαι θέση και να αποφασίζεις κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν βρούμε τίποτα χρήσιμο να προτείνουμε, θα συμφωνήσω κι εγώ. Η κατεξοδότηση πράξη τώρα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιούμε, αλλά να έχουμε και σωστή ε, συμπεριφορά και αντιμετώπιση ένα απέναντι στον άλλον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένω απαντήσει. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κράου από τη Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν αρκετά θέματα. Θα ήθελα να διευκρινίσω καταρχάς ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, άπτεται απλώς ε, συγκεκριμένων στοιχείων που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται στην ε, κείμενη, στον κείμενο κανονισμό επιτροπολογίας. Η πρόταση δεν αφορά τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση να ακολουθούν διαφορετική διαδικαστική οδό και αυτή εδώ απορρέει απευθεία από τη συνθήκη. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο τις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες απορρέουν από τον ε, κανονισμό για τις εκτελεστικές πράξεις του 2011. Και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει να αλλάξει εκ το πλαίσιο της επιτροπολογίας, αλλά προσπαθεί να απαντήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα πρόβλημα το οποίο βιώνει από το 2011 και μετά και αυτό είναι αυτό το οποίο πολύ σωστά ε, ανάφερα κάποια ε, ε, μέλη και αφορά την διαδικασία του έφεσης. Η διαδικασία της Επιτροπολογίας λειτουργεί πολύ καλά. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει περίπου 1.500 εκτελεστικές πράξεις το χρόνο. Περίπου 98% αυτών των πράξεων, των 1.500 ε, δηλαδή εκτελεστικών πράξεων, περνούν από ε, διαδικασίες επιτροπολογίες με θετική γνωμοδότηση από τα κράτη-μέλη. Ε, Σπανίω υπάρχουν αρνητικέ γνωμοδοτήσει και υπάρχει αυτό το 2% της, μη γνωμοδότησης. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα δηλαδή της γνωμοδότησης, δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών, είτε υπέρ είτε κατά μιας πρότασης και ε, βάσει κάποιων προϋποθέσεων και βάσει κάποιων εναλλακτικών εκδοχών, όπως για παράδειγμα αντίθεται θέμα ασφάλειας ε, ανθρώπων, ζώων και φυτών, το ε, θέμα πηγαίνει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην Επιτροπή Εξέτασης της Έφεσης. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αναφερθήκατε ήδη στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, ε, έχουμε το εξής. Δεν ε, είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο ήλπιζε ο κανονισμός επιτροπολογίας, δηλαδή να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε κάποια λύση. Τελικά δεν καταλήγουμε σε λύση και ουσιαστικά να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα της ε, Επιτροπής Επιτροπολογίας. Και αυτή φυσικά είναι μια κατάσταση που προκύπτει ακριβώς γιατί Αυτές ε, οι περιπτώσεις ε, είναι τόσο ευαίσθητες σε πολιτικό επίπεδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επιλύσει το πρόβλημα. Και ένα από τα μέλη το ανέφερε, ε, είναι λίγο ατυχές να πολιτικοποιούνται αυτές οι διαδικασίες. Δεν έχει κανένα συμφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πολιτικοποιήσει τις διαδικασίες. Ε, τα κράτη-μέλη σε αυτές τις περιπτώσεις ε, δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και προσπαθούν να ε, δώσουν το φλέγον θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποια πράγματα προκύπτουν απευθείας από τη βασική νομική πράξη, την οποία έχουν εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και για να μπορέσουν να έχουν ομοιόμορφους κανόνες εφαρμογής, έχουν εκχωρήσει κάποιες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ τα κράτη-μέλη διαδραματίζουν τον εξή ρόλο, ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην άσκηση αυτών των εξουσιών μέσω της Επιτροπής Επιτροπολογίας. Και ακριβώς ε, λόγω αυτής της εμπειρίας ε, τελικά έχουν ε, ξαναβρεθεί αυτά τα ζητήματα στην ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πέσει στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση, να αλλάξουν κάποια στοιχεία στη διαδικασία της Επιτροπολογίας, τέσσερα στοιχεία, κάποια από εσάς τα αναφέρατε ε, και εδώ και αυτό προτείνει στην ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις στο μέλλον υπό την προπόθεση βέβαια ότι θα γίνει αυτή η πρόταση από ε, λίγα κράτη-μέλη. Το αντίθετο ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα έχει αποτέλεσμα, απλώς ελπίζουμε να λειτουργήσει το σύστημα. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, νομίζω ότι τα ακούσαμε και από εσά και από άλλε επιτροπέ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που υποστηρίζουν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγαλύτερη διαφάνεια για τι ψήφου των ε, κρατών μελών και αυτό θα το υποστηρίξετε και εσεί από ό,τι ακούμε. Νομίζω ότι αρκούν αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε άλλε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής μας τώρα, ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους, αλλά ε, για όλα τα σχόλια που είναι ενδιαφέροντα και απαραίτητα. Όλοι κατανοούμε ε, το πρόβλημα, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και μία είναι η λύση. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να θα μπορούσε να είναι πιο ευνοϊκή στην άποψή της. Εμείς έχουμε κάποια αιτήματα για διαφάνεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ε, δύσκολα ζητήματα, για ευαίσθητα ζητήματα. Μας είναι πολύ προσφυλή αυτά τα θέματα. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε, τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας και ελπίζω να ε, συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μέχρι να βρεθεί μια κοινή λύση ικανοποιητική για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τους συναδέλφους για τη συζήτηση, τις απαντήσεις. Ε, μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου έχετε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. 7 Σεπτεμβρίου, μία το μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσει αύριο η Επιτροπή με την Προεδρία του κ. Ντεκάστρο. Εγώ σας αποχαιρετώ. Και ολοκληρώνουμε την απογευματινή συνεδρία. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Κύριε Σοδοπέρα, στις απογευματινή συνεδρία